So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Καλημέρα, συνάδελφοι. να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία δύο εκθέσεων και μετά έχουμε την συζήτηση του εργαστήριου για την πανδημία της γρήπης 1 Καταρχάς, να ψηφίσουμε την αναθεώρηση του σχεδίου δράση για την ενεργειακή απόδοση. Μια έκθεση της ε, Επιτροπής ε, Βιομηχανίας, γνωμοδότηση του κυρίου Λίζε. Έχετε μπροστά σας ε, τον κατάλογο ψηφοφοριών. Χθες το βράδυ προέκυψε και μια νέα έκδοση του καταλόγου. Ελπίζω να έχετε τη σωστή σας, τη σωστό, έγγραφο μπροστά σας. Έχετε λοιπόν και τις κάρτες μαζί, σε περίπτωση που χρειάζεται να ελέγξουμε. Ο κύριος Λίζα, διαδικαστικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξαφνικά φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον που επικρατεί για την γνωμοδότηση αυτή. Το συζητήσαμε με 5-6 άτομα στο Στρασβούργο και δεν υπήρχαν τότε πολλά αμφιλεγόμενα στοιχεία, αλλά ε, φαίνεται ότι είναι εκρηκτικό το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, γιατί απαιτούμε πάρα πολλά, δικαίως θεωρώ, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει χωρίς συζήτηση, φαντάζομαι. Η θέση λοιπόν της ε, Επιτροπής μας θα πρέπει να είναι σαφής, προκειμένου να το πετύχουμε αυτό με τους ε, σκιώδης, υπέβαλα τροπολογίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο τροπολογιών ψηφοφορίας και λυπάμαι που καθυστέρησα και σας τις υπέβαλα χθες το βράδυ. Νομίζω ότι πολλοί ξύπνησαν και κατάλαβαν πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις που κρύβονται στην γνωμοτότηση αυτή. Πέρα από αυτά που αναφέρονται στο κατάλογο ψηφοφορίας, θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. το σημείο 3 της αρχικής έκθεσης, για τους μακροπρόθεσμους στόχους της αρχικής έκθεσης, να τους ψηφίσουμε ξεχωριστά. Είναι πολύ φιλόδοξη αυτή η στόχη. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι και από πλευράς της Επιτροπής μας ιδιαίτερα σημαντική είναι η στόχη αυτή βασίζονται σε ένα σενάριο ότι θα υπάρχουν μόνο ανανεώσιμες ενέργειες το 2050 αλλά επικρατεί η άποψη ότι δεν θέλουμε 100% ανανεώσιμες ε, ε, ενέργειες, θέλουμε και άλλους τρόπους ενέργειας και θα πρέπει να προσαρμοστούν κάποια αριθμητικά στοιχεία. Εμένα αυτό που μου φαίνεται σημαντικό είναι να δώσουμε μία μακροπρόθεσμη προοπτική στη βιομηχανία προκειμένου να προσαρμοστεί σταδιακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συνεργασία σας. Να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους, το, τη γραμματεία που με βοήθησαν τόσο πολύ χτες το βράδυ και τους συναδέλφους τους και όλους εισηγητές και να σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί ήταν επιτακτική ανάγκη να, βάλουμε κάποιες τροπολογίες κοιτώντας την ε, τροπολογία 40 για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Έλαβα από περιβαλλοντικές ενώσεις ε, ένα email το οποίο ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένη η ημερομηνία το 2050 για να έχουμε προσαρμόσει τα κτίρια ενώ άλλοι συνάδελφοι από ομάδε άλλε μου παρατήρησαν ότι ήταν ακριβώ πάρα πολύ νωρί. Το αντίθετο δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται συζήτηση για να δούμε κατά πόσο είναι το 2040, το 2050 η κατάλληλη ημερομηνία. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος να δούμε, να αποφασίσουμε ποια είναι η πιο κατάλληλη ημερομηνία. Να περάσουμε στην τροπολογία 1 της Κατλέν Φαμπρέντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Σκυλακάκης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 5. Υπέρ. Κατά.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 Άποχες. Απορρίπτεται. Η 14 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 15 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται Η 40 με προφορική τροπολογία. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 38 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 39 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 18 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Αν το ελέγξουμε παρακαλώ. Για 18. Πέρα ψηφοφορία. 28. υπέρ, 25 κατά εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, 23 υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. Η 30 υπέρ. Η 24, συγγνώμη, δεν λοιπόν, πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η 17. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. άποχε. Εγκρίνεται. Η 37 σε τμήματα. Πρώτο το τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. EPP Από το ΕΛΚ ψηφίζει ένας παραπάνω, παρακαλώ. Ist gut. Εντάξει. Απορρίπτεται. Η 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 35 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 27 αποσύρθηκε. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 36 υπέρ. Και αυτή εγκρίνεται. Και περνάμε ηλεκτρονικά στην τελική ψηφοφορία. Έναξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρασε. 46 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, μία αποχή. Να συγχαρούμε τον εισηγητή, τον κύριο Πέτερ Λίζα. Σημαντικό το θέμα αυτό, το οποίο το ακούσαμε και χτες από την Επίτροπο για την αλλαγή του κλίματος. Συγχαρητήρια. Der Punkt 10 COP16. Το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, το 10, COP16. Διάσκεψη των Ηνωμένων Αθηνών για το κλίμα στο Κανκούν. Σεπτεμβρίου ήταν η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Μεγάλο ο κατάλογο ψηφοφοριών. Να ξεκινήσουμε. Η ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η δύο υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Η τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 18 και η 30 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να συνεχίσουμε. Η 20 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. ελέγξουμε την 25, λέει ο Πρόεδρος, ηλεκτρονικά. Abstimmung beendet. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν 24, έχει αποσυρθεί 28, 26 λοιπόν τώρα, του κυρίου Φλόρεντς υπέρ. Κατά. Άποχες Εγκρίνεται 29 και 27 που είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 30 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 33. Συγγνώμη, είναι 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 35. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η παράγραφος 5 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Η 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είσαι 54 και η 57 που είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε για την 54-57. Ε, Πάλι περισσεύει ένας από το ΕΛΚ και ένας από τους σοσιαλιστές. Από τους σοσιαλιστέ ακόμα ένας. Jetzt ist gut. Εντάξει τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 54 και 53 που είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 73 και οι 72 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 65 ist Beendet. Εγκρίνεται. 62 fällt. 62. 60 σκυλακάκες. 66 σκυλακάκες. Να ψηφίσουμε παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην επόμενη σελίδα περνάμε τώρα. Στην 64. Υπέρ. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 74 είναι γλωσσικής φύσεως. 88 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 56 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 90 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 59 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε για την 59. Ein PP zu viel. Jetzt ist gut, beendet. Πέρας. Εγκρίνεται. Για την 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 84 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Η 80 και η 81 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83-77 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86-87 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές Α, συγγνώμη, άλλη μια φορά για την 85 παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 91 Β και η 92 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η ΔΕΒΕ 96 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό εγκρίνεται. Και τώρα λοιπόν η 116. Παρνιό. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, υπορρίπτεται, συγγνώμη. Καταπίπτει 102 ή 100. Πρέπει να τις ψηφίσουμε. Την 102, παρακαλώ, υπέρ. Φαν την 102, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η 100, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 101. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 103 με σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Abstimmung beendet. Πέρασε. Ja, abgelehnt, ne? Ναι, όντως απορρίπτεται. Καταπίπτει 97 και έτσι περνάμε στην 97 δεύτερο τμήμα. Part B, υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές ε, γκρίνεται η 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 107 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Ταυτόσιμες. Οι 110 και οι 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν έντεκα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 106. Καταπίπτει. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 113 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα. Und beendet. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε για την 114. Πέρασε. Πέρας. Απορρίπτεται. 115. Φλόρεντς Ιμπερλίδη. Υπέρ. Εκατόν δεκατέσσερα την ψηφίσαμε. Και τώρα περάσαμε στην 115, λέει ο πρόεδρος. Ψηφίσαμε ηλεκτρονικά τον 114, απορρίφθηκε, λέει ο πρόεδρο. Συγγνώμη, συγγνώμη, λάθο, Βιάστηκα. 114, λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν. 115 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύε 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Για την 119. Abstimmung beendet. Πέρας. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ 126 να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορία. Ja, Abstimmung ist Εγκρίνεται. Stimmt aber auch nicht jeder mit Αλλά δεν ψηφίζουν όλοι με κάρτα. Γι' αυτό λοιπόν κάπως μπερδευόμαστε. 110... 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 στα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 ντεβε σε τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται 137 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται 157 καταπίπτει και περνάμε στην 139 στα τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 144. Part B. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 part A. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180... 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 153. Ηλεκτρονικά. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Γι' αυτό δυσκολεύομαι. Εγκρίνεται. Η 153 εγκρίνεται. 154 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 155. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 154. Εντάξει. EPP ε, Ανατσεφίλ. Περισσεύει από το ΕΛΚ. Εγκρίνεται. 155 της Ήπρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 197 κατά αποχές απορρίπτεται 156 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 part B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 μερικής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 λέει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 159 Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 160 στα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά. Άποχες τα 182 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 182. Abstimmung beendet. Πέρασε. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 162 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 τη ίδιες σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα. Abstimmung beendet. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εκατόν εξήντα υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 165. Beendet. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 170 Abstimmung beendet. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 167 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 173 και 174 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120, συγγνώμη. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε για την 124 με προφορική τροπολογία, παρακαλώ. ist beendet. Πέρας. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν εννέα υπέρ. Γκαρντίνι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε μου λένε ότι έχουν διαγραφεί δύο τροπολογίες. Η κυρία Σούλη και ο κύριος Φράνκο δεν υποστηρίζουν την τροπολογία. Θα την ψηφίσουμε, αλλά χωρίς τα δύο ονόματα αυτά. Η 200 part B υπέρ. Η 200 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες Απορρίπτεται. 204 γκαρντίνι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ. Ναι, χωρίς τα δύο ονόματα. Τα υπόλοιπα διατηρούνται. Υπέρ λοιπόν για την 202. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 203. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 206 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 209 και η 207 και οι 47 που είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 210. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στι ιδεολογικές σκέψεις. 6. Δελβό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9. Υπέρ. Συγγνώμη, η 8. Στην 8, στην 8 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Για την 8. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την εννέα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η δέκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. οι 14 στα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της 14 παρακαλώ. Abstimmung beendet. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Η 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και τώρα να κάνουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Ein PPP zu viel. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚΑ. Πέρας ψηφοφορίας. 35 ψήφοι υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή. Να συγχαρούμε λοιπόν τους εισηγητές της έκθεσης αυτής που θα αποτελέσει μια σημαντική βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις μας μέχρι την Ολομέλεια και μέχρι την ε, συνδιάσκεψη στο Κανκούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο εργαστήρι για την πανδημία της γρήπης. time. I, Please take a seat. Καθίστε παρακαλώ. So, herzlich willkommen an alle Mitglieder des Ausschusses. Να καλωσορίσω όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής μας και όλους τους εμπεριογνώμονες καθώς και όλους τους προσκαλεσμένους μας στο εργαστήριο αυτό για την ε, διάσημη γρήπη ή τα ένα με την οποία ασχοληθήκαμε τόσο εντατικά πέρσι. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε τις αντιδράσεις των κρατών μελών και τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τον εισηγητή, την εισηγήτρια η οποία θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό, το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ έντονε και δραματικές ε, δημόσιες αντιδράσεις. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας μία σειρά εμπρογνωμόνων, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει εν μέρη. και είχαν διαδραματίσει διαθεσμικό θεσμικό συγγνώμη ρόλο. Καλωσορίζω και με τη σειρά που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Τον κύριο Τζον Εφράιαν, ο οποίος είναι από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, επικεφαλής. Στη συνέχεια και πάλι από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ έχουμε τον κύριο Άντρεϊ Ρίς, ο οποίος είναι Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων. Μετά έχουμε την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων Enterprise με την κυρία Ζορζέτ Λαλή, η οποία είναι επικεφαλής της βιομηχανικής καινοτομίας και των βιομηχανιών κινητικότητας. Από την προηγούμενη Σουηδική Προεδρία έχουμε μαζί μας την κυρία Ανίτα Γιανέλμ. Σας καλωσορίζουμε. Η Σουηδική Προεδρία αντιμετώπισε σε μεγάλο μέρος ε, την ιστορία αυτή. Χαίρομαι ε, επίσης που έχουμε μαζί μας τον Executive Director της ΕΜΑ, τον κύριο Τόμας Λουντρεν. Καλώς ήρθατε. Και τέλος την ε, πρώην Διευθύντρια του ECDC, την κυρία Σουζάνα Γιακάμπ. Έχουμε φυσικά μαζί μας και τον τρέχον επικεφαλής του ECDC, τον κύριο Σπρέγγερ. Σας ε, καλωσορίζουμε και εσά, κύριε Σπρέγγερ. Και άλλου δύο προσκεκλημένους μαζί μα από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, την Γενική Διευθύντρια Παόλα Τεστορικότσι. Καλώ ήλθατε και από την Βελγική Προεδρία, τον κύριο, τον δόκτωρ Ντάνιλ Ράιντερ. Δεν ε, τήρησα το πρωτόκολλο, απλά διάβασα τα ονόματα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Όπως είπα, ήταν μεγάλη ταραχή που επικράτησε πέρσι για τον ιό αυτό. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η οποία είχε προβλέψει μια πανδημία, προκάλεσε αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ευτυχώς τα πράγματα δεν εξελιχθήκαν όπως φοβούνταν, πολύ. Και τώρα τίθεται μια σειρά ερωτημάτων για το πώς ε, μπορούμε να οργανώσουμε την αντίδρασή μας σε τέτοιους ιούς, σε τέτοιες απειλές διακρατικής φύσεως. Και γι' αυτό λοιπόν ε, διοργανώσαμε το σημερινό εργαστήριο. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια χρονικά περιθώρια. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 12.30 το οποίο μπορεί να ακούγεται πολύ, αλλά δεν είναι πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ο κάθε ομιλητή θα πρέπει να τηρήσει χρονικό περιορισμό. Ο κύριος Τζον Ράιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 λεπτά και οι υπόλοιποι ε, ομιλητές 4 λεπτά. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Ράιαν να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Thank you very much, Mr. Chair. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για τη διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου μαζί με την συνδιάσκεψη της Βελγικής Προεδρίας για τον ιό H1N1 που έγινε τον Ιούλιο και μαζί με άλλες συναντήσεις που έχουν γίνει για το ζήτημα αυτό, ελπίζω ότι και το σημερινό εργαστήρι θα βοηθήσει στο να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση. Έχουμε αποκομίσει κάποια πολύ σημαντικά διδάγματα από την πανδημία αυτή της γρήπης και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο στο μέλλον να βελτιώσουμε την ανταπόκρισή μας και την αντίδρασή μας σε τέτοιες κρίσεις υγειονομικές και να προστεύσουμε καλύτερα τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς να συνειδητοποιήσουμε το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτιλήθηκε η όλη προετοιμασία της ετοιμότητας και της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία της γρήπης και θα ήθελα ακριβώς αυτό να αφαιρθώ στη δική μου παρουσίαση από το 1999 προκειμένου να αντιμετωπίσουμε απειλές που είχαν να κάνουν με ε, μεταδοτικές ασθένειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην έγκριση κάποιων νομοθετικών πράξεων. Βασικός στόχος των νομοθεσιών αυτών ήταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού της δράσης που λαμβανόταν κατά των μεταδοτικών ασθενειών συμπεριλαμβανομένης της γρήπης. Ενδυναμώθηκε η στρατηγική αυτή το 2005 όταν εγκρίθηκε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της πανδημικής γρήπης που είχε ως στόχο να συντονιστούν καλύτερα τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των κρατών μελών. Επίσης δημιουργήσαμε ανεξάρτητους οργανισμούς με εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως για παράδειγμα η ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ελέγχου Νόσων και η ΕΜΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Παρ' όλα αυτά δεν προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη καμία διάταξη για την αρμόνιση της ε, εθνικής πολιτικής δημόσιας υγείας των κρατών μελών. Μόνο η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται σε κάποια μέτρα διασυνοριακής αντιμετώπισης απειλών στη δημόσια υγεία. Εν συντομή θα μπορούσε να πει κανεί ότι η βασική ευθύνη αντιμετώπιση των κρίσεων απόκειται ακόμα μόνο στα κράτη-μέλη, ότι σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχει κάποιος συντονιστικός ρόλος. Θα ήθελα πολύ σύντομα να δούμε κάποιε βασικέ ημερομηνίε όσον αφορά την εκδήλωση τη πανδημία. Καταρχά, με διμερείς επαφές που είχαμε με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, συνειδητοποίησαμε ότι είχε εμφανιστεί ο νέος ιός. E Αυτό σύντομα επιβεβαιώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ελέγχου των Νόσων δραστηριοποιήθηκε και ζήτησε άμεσα από τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εξετάζουν την κατάσταση της δημόσιας υγείας και να αρχίσουν να σκέφτονται τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της νόσου. Γινόντουσαν στη συνέχεια συναντήσεις σε καθημερινό επίπεδο προκειμένου να, μπορούν να, προκειμένου να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τη μετάδοση της νόσου και προκειμένου να, να μπορέσει να ληφθεί η κατάλληλη δράση για τον περιορισμό της νόσου. Στα πρώτα στάδια της μετάδοσης ε, του ιού τα κράτη-μέλη εξέτασαν τη δράση που θα μπορούσε να ληφθεί ιδίως όσον αφορά τους ταξιδιώτες οι οποίοι ε, φτάνανε ή ερχόντουσαν από περιοχές ε, επικίνδυνες. Επίσης εξέταζαν τις συμβουλές που θα μπορούσαν να δώσουν προληπτικά στους ε, μελλοντικούς ταξιδιώτες. Για παράδειγμα κάποια βασικά μέτρα υγιεινής ή η χρησιμοποίηση κάποιων αντιοικών φαρμάκων όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια ένα δεσμευτικό ορισμό των ε, κρουσμάτων πράγμα το οποίο οδήγησε στη θέσπιση ενός ε, συστήματος παρακολούθησης της μετάδοσης του ιού στα πλαίσια της κοινότητας. Στις 11 Ιουνίου του 2009, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέβασε το επίπεδο συναγερμού για την πανδημία στο επίπεδο 6. Πρώτη φορά λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο παγκόσμιας πανδημίας. Μετά τις ε, πάρα πολλές συναφορές που είχαμε για την εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη, καθώς επίσης και μετά την ακίνωση των πρώτων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας προχώρησε στην υποβολή συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να υπάρχουν πλέον κοινά μέτρα και κοινέ αρχές για την μετώπιση της νόσου. Γίνανε κάποιες δηλώσεις όσον αφορά το κλείσιμο των σχολείων, καθώς επίσης και όσον αφορά την θεραπεία και τη μετώπιση των ασθενών. Επίσης, η Επιτροπή Ασφάλεια τη Υγεία έκανε κάποιε συστάσεις όσον αφορά τη στρατηγική εμβολιασμού, δηλαδή ποιοι τομεί του πληθυσμού θα έπρεπε να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια δημοσίευσε το Σεπτέμβριο του 2009 μία ανακοίνωση όσον αφορά την πανδημία της γρήπης με πέντε συγκεκριμένα έγγραφα που είχαν να κάνουν με βασικά ζητήματα της διαχείρισης και της αντιμετώπισης της κρίσης. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2009 μετά από κάποιες θετικές συστάσεις από την υπηρεσία φαρμάκων για την ανθρώπινη χρήση, ξεκίνησαν τον Οκτώβριο συγκεκριμένα οι πρώτες εκστρατείες εμβολιασμού. Το ζήτημα αυτό δεν θα αναπτυχθεί περισσότερο από τις επόμενες παρεμβάσεις. Ορισμένα κράτη-μέλη δήλωσαν ότι ήδη είχαν κάνει σημαντικές παραγγελίες για εμβόλια, αλλά πάλι όχι προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, το δεν υπήρχε δηλαδή κάποια συντονισμένη δράση ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε στα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν ε, τις ε, διαδικασίες παραγγελίας των εμβολίων. Επίσης, αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε ένα σύστημα μεταφοράς κάποιων εμβολίων από τη μία χώρα στην άλλη, από τις, από τις χώρες που είχαν εμβόλια σε αυτές οι οποίες δεν είχαν αρκετά εμβόλια. Επίσης, ε, πολύ σημαντικά κρούσματα είδαμε και στην ε, Βουλγαρία, καθότι όχι μόνο δεν υπήρχαν εμβόλια στη χώρα αυτή, αλλά ούτε και τα απαραίτητα αντιϊκά φάρμακα. Επίσης, στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας υπήρχε ο κατάλληλος συντονισμός, αλλά παράλληλα τα απαραίτητα Συμβούλια Υπουργών Υγείας, τα αρμόδια Συμβούλια Υπουργών Υγείας συνεδρίαζαν πολύ συχνά προκειμένου να συντονίσουν εθνική δράση. Επίσης, κλήθηκαν οι χώρες του G7 μαζί με το Μεξικό να προχωρήσουν σε έναν καλύτερο συντονισμό της αντιμετώπισης της γρήπης προκειμένου να βοηθηθούν καλύτερα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 ξεκίνησε μία αξιολόγηση της ε, αντιμετώπισης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία της γρήπης. Στόχος αξιολόγησης αυτής ήταν να καταφέρουμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από την εκδήλωση της πανδημίας αυτής και προκειμένου κατά αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων της δημόσιας υγείας. Έχουμε προχωρήσει συγκεκριμένα στη δημοσίευση δύο εκθέσεων, οι οποίες θα υποβληθούν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμπληρωθούν οι εκθέσεις αυτές από τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιήσει η Βελγική Προεδρία μετά την ε, συνεδρίαση που διοργάνωσε τον Ιούλιο και βέβαια στα συμπεράσματα αυτά θα συμβάλλουν και τα πορίσματα του σημερινού εργαστηρίου. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή άντλησης διδαγμάτων από την πανδημία και ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε και προκειμένου να ξεκινήσει και η συζήτηση Όσον αφορά την αξιολόγηση της ε, αντίδρασή μα, ανταπόκρισής μας, θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποιες βασικές αποφάσει που ελήφθησαν σε κοινοτικό επίπεδο. Καταρχάς, το case definition, να καταφέρουμε δηλαδή να ορίσουμε τι σημαίνει κρούσμα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να αντιμετωπίσουν γρήγορα και συντονισμένα την εκδήλωση της γρήπης. Επίσης, προκειμένου να έχουμε την απαραίτητη πολιτική δέσμευση, τα κράτη-μέλη ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που ζητούσαν για περισσότερο συντονισμό και αλληλεγγύη στη διαχείριση της κρίσης. Τρίτον, η πολιτική αυτή δέσμευση εφαρμόστηκε πολύ περισσότερο μέσω δηλώσεων και συστάσεων όσον αφορά τη διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου μέσω της Health Security Committee της Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση στη συνέχεια και πέντε έγγραφα εργασία το Σεπτέμβριο που αναφέρονταν στα σημαντικότερα σημεία της διαχείρισης της κρίσης. Η όλη αυτή η εργασία καθώς επίσης και οι πρωτοβουλίες βασίζονταν στις βασικές επενδύσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της τα τελευταία αυτά χρόνια στην βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε και σαφώς πολύ περισσότερα πράγματα πρέπει να συμβούν στο μέλλον για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Ελπίζω ότι οι εκθέσεις και εξορρογήσεις στις οποίες αναφέρθηκα καθώς επίσης και το σημερινό εργαστήρι θα βοηθήσουν να βελτιώσουμε το σύστημα τιμότητας που έχουμε για να προσθέσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τώρα τέσσερι πιναλίστε μαζί μα οι οποίοι θα απαντήσουν τα τρία ερωτήματα που θέσαμε. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Αντρέ Ρίς από την Γενική Διεύθυνση Σάνκο να μας απαντήσει σε τέσσερα λεπτά. Uh, thank you very much, uh, Members. Uh, σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου. Ακούσατε στην προηγούμενη παρουσίαση ποια ήταν τα βασικά σημεία ανταπόκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία. Προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα το σύστημα αυτό αντίδρασης, ανταπόκρισης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια ήταν τα βασικά σημεία που διέπουν την προσπάθεια που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταπόκριση αυτή είχε ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη λειτουργούσαν με τρόπο συντονισμένο βάσει των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων. Και όπως είπε και ο κύριος Ράιαν, ο συντονισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέτρο, ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο στη συζήτηση που κάνουμε. Επίσης θελήσαμε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας αυτής στην κοινωνία καθώς επίσης και στη λειτουργία των επιχειρήσεων του οικονομικού τομέα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτα έτοιμος για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Ωστόσο, με την κατάλληλη προετοιμασία και τον κατάλληλο στονισμό, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές μπορούν να βοηθήσουν στο να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις μιας πανδημίας. Και πιστεύω στεναρά ότι κατά τη διάρκεια τη δημόσια αυτή ε, κρίση μιας τόσο σημαντικής κρίσης δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, η πρώτη μάλιστα τέτοια, είναι μια περίπτωση που κατέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει πολύ καλά την κρίση αυτή, ενώ είδαμε ότι σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως στην Ουκρανία, η ετοιμότητα αυτή δεν υπήρχε. Αρχικά, η αρχές του Μεξικού ήρθαν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάφερε κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να αντιμετωπίζει καλύτερα την κρίση σε διασυνοριακό επίπεδο, κατάφερε να πετύχει τον κατάλληλο συντονισμό σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί έξι εξασφαλίσαμε μια πολύ καλή συνεργασία στην ανταπόκρισή μας. Θα ήθελα να σας πω ότι εξ αρχής είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, η Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η Γενική Διεύθυνση για τα Εμβόλια και τα Φαρμακευτικά Προϊόντα συνεργάστηκαν πολύ αποτελεσματικά και δημιούργησαν τον μηχανισμό αυτών που μας επέτρεψε να καταφέρουμε να πετύχουμε τον κατάλληλο στονισμό και στο εσωτερικό των κρατών αλλά και διασυνοριακά. Επίσης προχωρήσαμε στα πολύ καλό σύστημα ανακοινώσεων. Σε καθημερινό επίπεδο εκδίδαμε ανακοινώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες πήγαιναν προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ε, Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας, η Health Security Committee, ήταν η αρμόδια για το στονισμό της δράσης των κρατών μελών. Η Health Security Committee έδινε τις απαραίτητες συστάσεις τόσο για τους ταξιδιώτες όσο και την ε, εκστρατή εμβολιασμού των κρατών μελών. Βάσει των προτάσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά την έγκριση των δηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη-μέλη είχαν αρχίσει να υιοθετούν συνεκτικά συνεπίπλεον μέτρα συντονισμένα μεταξύ τους. Η θέση πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Και θα ήθελα να σας πω επίσης ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ε, πανδημίας και νέκρινε κάποιες ε, πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα το σωστό σύστημα υποβολής αναφορών για την παρακολούθηση της ε, πανδημίας και για την έκδοση των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων. Ο πρόεδρος Γιακόπ, νομιλητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο συγκεκριμένε υπηρεσίε που μα υποστήριξαν, την ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη Ελέγχου των Νόσων. Ο πρόεδρο διακόπτει μιλητή. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Κυρία Λαλή, έχετε το λόγο. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν υπεύθυνη για την έγκριση στην αγορά του εμβολίου, τότε που ανακηρύχθηκε η πανδημία, τότε που η Γενική Διεύθυνση Enterprise ήταν υπεύθυνη για τα ιατρικά θέματα, για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Θα σας αναφέρω λοιπόν τι συνέβη μέχρι τον Φεβρουάριο 2010, τότε που το, ο φάκελος αυτός μεταφέρθηκε στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Το 2005 όταν ε, υιοθετήθηκε το σχέδιο ετοιμότητας για την πανδημία δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για να διατεθεί επιγόντως ε, ένα τέτοιο εμβόλιο όπως τότε που χρειάστηκε ε, για την πανδημία της γρήπης με επίπεδο 6. Μετά την μεταρρύθμιση του 2004 είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια και χρειάστηκε λοιπόν ένα νομικό πλαίσιο να προετοιμαστεί για να δοθεί άδεια διάθεση στην αγορά στο υφιστάμενο πλαίσιο του 2005. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι το εμβόλιο για την πανδημία αποτέλεσε μια εκδοχή της εποχιακής γρήπης και των σχετικών εμβολιασμών. Γι' αυτό λοιπόν χρειάστηκε να υπάρξει ένα ένας φάκελος βασικός φάκελος και το 2009, τον Ιούνιο του 2009 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, ανέβασε το επίπεδο κινδύνου στο επίπεδο 6 χωρίς ε, να έχουμε τα κλινικά στοιχεία. Ακολουθήσαμε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ωστόσο, εντός των ε, νόμιμων, των νομικών ε, προδιαγραφών, κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε συνδυασμό και σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ σπρώξαμε όσο μπορούσαμε αυτά που μας έδωσαν ε, οι επιστήμονές μας. Τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας μεταξύ Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου έγιναν κλινικές ε, δοκιμές στο νότιο ημισφαίριο, οι οποίες και δεν ε, ολοκληρώθηκαν. Γι' αυτό ήταν υπό όρους οι αδιαδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι προσπαθήσαμε να ασκήσουμε πίεση και η υπηρεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σπρώξαμε στα άκρα σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα των στοιχείων. Οι βασικές ομάδες κινδύνου ήταν οι έγκυες και τα νεαρά παιδιά. Για, τα, για τις οποίες δύο ομάδες είχαμε και τα πιο περιορισμένα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν καταφέραμε να διαθέσουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα, δια, ήταν στη διάθεση της Ευρώπης από την αρχή του χειμώνα, το οποίο θα πληρούσε τις προδιαγραφές ασφαλείας και νομίζω ότι πραγματικά καταφέραμε να ανταποκριθούμε στα δύο βασικά προβλήματα που ήταν η ετοιμότητα και η προστασία. Ευχαριστώ κυρία Λαλής, λέει ο πρόεδρος και τώρα περνάμε στην ε, πρώην Σουηδική Προεδρία, στην κυρία Γιαννέλμ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στο εργαστήριο αυτό. Ε, καλέσατε την Υπουργό μας, αλλά λόγω της ανακοίνωσης της νέας κυβέρνησης της Σουηδία σήμερα δεν μπόρεσε να προβλεφθεί σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα την εκπροσωπήσω. Καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά διστακτικοί και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την εξαγωγή τελικών πορισμάτων. Κατά δεύτερον, η λήψη αποφάσεων κατά, την, ε, κατά τη ε, διάρκεια κρίσεων πάντα γίνεται υποπίεση χωρίς να έχουμε επαρκή στοιχεία, αλλά δεν έχουμε την ε, πολυτέλεια να μην λαμβάνουμε αποφάσεις κατά τη διάρκεια κρίσεων και θα πρέπει φυσικά οι αποφάσεις να λαμβάνονται υπό, να, να λαμβάνονται παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην επαρκούν τα επιστημονικά στοιχεία, γιατί είναι πιο καλό να λαμβάνονται αποφάσεις από το να μην λαμβάνονται. Πρέπει να αναλαμβάνεται δράση σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, όπως είπε και ο Τζον Ράιαν, ότι πρόκειται για έναν τομέα με μεγάλη αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία είναι αρμόδια σε επιχειρησιακό επίπεδο, ότι το επίπεδο δράσης που λαμβάνεται εναπόκειται στα κρατημέλη και ότι οι πιο πολλές παρεμβάσεις λαμβάνονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και επίσης μια βασική αρχή για τις κρίσεις είναι ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα άτομα που πλήττονται από την κρίση. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν συντονίσαμε, ότι δεν συνεργαστήκαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κάναμε αυτό. Και θεωρούμε ότι το κάνουμε με επιτυχία. Τι έγινε λοιπόν υπό τη Σουηδική Προεδρία. Έγινε μια διάσκεψη εμπειρογνώμων τον Ιούλιο, ανεπίσημη υπουργική συνάντηση μετά από το συνέδριο αυτό και συζητήθηκε η πανδημία από τους υπουργούς. Στο Συμβούλιο επίσης έγιναν συζητήσεις. Ε, ε, επιπλέον υπουργική διάσκεψη έγινε για να συζητηθούν τα πορίσματα και χρησιμοποιήσαμε ασφαλώς ε, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετοιμότητα για την πανδημία. Ήταν καλή λοιπόν συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε συζήτηση το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, τελική συζήτηση και οι υπουργοί μας ε, ε, ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την υγεία. Τι πετύχαμε τον Ιούλιο στην διάσκεψη των εμπειρογνωμόνων. Ήταν ομόφωνη η απόφαση των κρατών μελών ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε τη στρατηγική μας και να περάσουμε σε μία στρατηγική περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας. Ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση. Επίσης, οι εμπειρογνώμονες αποφάσισαν ότι θα, θα έπρεπε να αναθεωρηθούν τα εθνικά σχέδια δράσης. Αλλά να θυμόμαστε ότι σε εποχές κρίσης δεν θα πρέπει να γίνονται πολλά, πολλές αλλαγές στα σχέδια ετοιμότητας Τέτοιε αλλάγέ θα πρέπει να γίνονται μετά τις πανδημίες και αυτό είναι βασικό σε ό,τι αφορά την αντίδραση και την ανταπόκριση σε κρίσεις. Επίσης, ε, τότε, τον Ιούλιο, συνειδητοποιήσαμε ότι κάποια κρατημέλη είχαν ε, συμφωνίες για τον εμβολιασμό, ενώ κάποια άλλα δεν είχαν σχετικέ συμφωνίες. Θα έπρεπε λοιπόν να αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον θέλαμε να υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα για την ε, παροχή, την προμήθεια των εμβολίων και κατά πόσον θέλαμε να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών των εμβολίων. Τα κράτη-μέλη επίσης ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει ενδεχόμενου ε, μελλοντικού ε, μηχανισμούς ε, για πρωτοβουλίες συνεργασίες. Όπω είπε και ο δόκτωρ Ράιαν. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αλλά Ίσως το Συμβούλιο θα μπορούσε να έχει τον ίδιο χρόνο όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπάμαι, δεν προβλέπετε. Θα επανέλθουμε, λέει ο Πρόεδρος μετά τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Να ζητήσουμε από τον κύριο Τόμας Λέγκριν να μας μιλήσει. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να απαντήσω στις τρεις ερωτήσεις που έχετε θέσει. Θα ξεκινήσω με την πρώτη. Ο ρόλος της ε, EMA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ήταν ο εξής. Πρόσβαση στα εμβόλια στο δυνατόν γρηγορότερα. Δεύτερον, η παροχή απαραίτητων πληροφοριών στους γιατρούς και τους ασθενείς. Και τρίτον, παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων από την στιγμή που είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς. Το 2003 είχαμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήμασταν έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημικής ε, κρίσης. Χρησιμοποιήσαμε ένα πολύ μεγάλο στόκ εμβολίων προκειμένου αυτά να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά την έγκριση του βασικού φακέλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρχίσαμε να κάνουμε τρεις δοκιμές ξεχωριστές προκειμένου να καταλήξουμε στο εμβόλιο από τη στιγμή που είχαν απομονώσει το στέλεχος του ιού της γρήπης. Η βασική μας στρατηγική εστέφθη με επιτυχία και αυτό φάνηκε και στη χρήση του εμβολίου που ακολούθησε στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά τον κίνδυνο, τη δεύτερη ερώτησή σας, βασιζόμαστε σε μια εμπειρία που έχουμε με την ε, εποχική γρήπη και με διάφορα στελέχη της εποχικής γρήπης. Κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση της ασθένειας κάθε φορά προτού προχωρήσουμε σε στρατηγική εμβολιασμού. Βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα, καθώς επίσης και στην ε, ιατρική πυρογνωμοσύνη. Είχαμε τρία συγκεκριμένα εμβόλια, τα οποία ήδη από την αρχή, από τις πρώτες δοκιμές που είχαμε κάνει, είχαν δείξει ότι μπορούσαν να λειτουργήσουν και ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος των ε, ασθενών, στους οποίους έγιναν οι δοκιμές. Επίσης η κατασκευαστική διαδικασία ήταν ε, πάρα πολύ καλή και είχαμε και την πολύ καλή συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών προκειμένου το εμβόλιο να μπορεί να διοχετευθεί, στους ασθενείς ε, στα πλαίσια πολύ αντίξεων και δύσκολων συνθήκων. Σήμερα περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί από το εμβόλιο αυτό της γρήπης και παρακολουθούμε συστηματικά την κατάσταση και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις από τα εμβόλια αυτά ή κάποιες συνεπιθύμητες παρενέργειες από τα εμβόλια αυτά. Περνά τώρα στο τρίτο σας ερώτημα. Το σχέδιο ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας επέτρεψε να έχουμε άμεσα την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη που υπήρχε σε κοινοτικό επίπεδο. Επίσης, στο, στην ισοσελίδα της ΕΜΑ του ε, Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Φάρμακα είχαν δημοσιευθεί απαραίτητες δηλώσεις για τις εκστρατείες εμβολιασμού καθώς επίσης και όλοι οι εμπειρογνώμονες με τα νόματά τους ήταν διαθέσιμοι στην ισοσελίδα αυτή. Οι συστάσεις που κάνει ο οργανισμός μας γίνονται κατά τον τρόπο που γίνονται και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε δηλαδή ένα συγητή, έχουμε εμπειρογνώμονες, κάθε μελέτη ε, εξετάζεται από ομότιμους και στο τέλος ε, καταλήγουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα, σε μια τελική σύσταση, ε, η οποία είναι απόλυτα αντικειμενική και δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα κανενός από τα συμβαλόμενα μέρη, από τους συντάκτες δηλαδή μιας έκθεσης. Επίσης υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στα πλαίσια της ΕΜΑ που δίνει πληροφορίες ακριβώς για την γρήπη. Θεωρώ λοιπόν τη διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν πέρα για πέρα για διαφανής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σουζάνα Γιάκαμπ η οποία ήταν πρώην διευθύντρια της ε, ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Ελέγχου των Όσων. Τώρα εργάζεται για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι θέλω να εργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην θέση που έχω, δηλαδή ως Περιφερειακή Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς ενέργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας της γρήπης. Θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα ήταν ήδη πολύ καλά σχεδιασμένα προτού εκδηλωθεί η κρίση, παρόλα αυτά μπορούμε να αντλήσουμε πολλά θετικά μαθήματα για να βελτιώσουμε τη στάση μας. Όταν ανέλαβα εγώ ε, τη θέση μου ως διευθύντρια του ECDC την 1η Μαρτίου 2005, το ECDC ήδη υπήρχε. Χρειάστηκε πολύ γρήγορα όμως να συντονίσουμε τη δράση μας και να αρχίσουμε να καταλήγουμε σε κάποιες πρώτες μελέτες και κάποια πρώτα πορίσματα. Ακόμα θυμάμαι ότι ε, ο τότε Επίτροπος ε, Κυπριανού είχε πάει σε κάθε κράτος μέλος προκειμένου να παρακολουθήσει την κατάρτιση των προγραμμάτων, των εθνικών προγραμμάτων ετοιμότητας. Αρχίσαμε να εργαζόμαστε για τα προγράμματα αυτά, τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα σε τρία χρόνια και συνέβαλαν πάρα πολύ στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πιο καλά προετοιμασμένη περιφέρεια προκειμένου να αντιμετωπίσει την πανδημία γρήπη. Το δεύτερο μήνυμα το οποίο θα θέλω να σα ε, αποστείλω είναι ότι το ευρωπαϊκό, το κοινοτικό σύστημα αλλά και το ECDC βασιζόταν στην τότε κοινοτική νομοθεσία για την ετοιμότητα και την ε, αντίδραση. Χρειάστηκε να συνεργαστούμε λοιπόν πάρα πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και με τις εκάστοτε προεδρίες και πρέπει να πω ότι η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της γρήπης. Χρειάστηκε να στήσουμε, όπως σας είπα, την ECDC πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλήξαμε πολύ γρήγορα και σε αποτελέσματα καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολλές αξιολογήσεις κινδύνου ήδη από το 2005 και όλο και περισσότερες καθώς εκδηλωνόταν η γρήπη. Όλες αυτές οι αξιολογήσεις κινδύνου ήταν ε, εντελώς ανεξάρτητες Υπογραμμίζω τη λέξη ανεξάρτητε, γινόντουσαν από του καλύτερου εμπειρογνώμονες που έχουμε, ήταν απόλυτα ισορροπημένε και απόλυτα διαφανεί και χρησιμοποιούσαμε αυτέ τι αξιολογήσεις κινδύνου στα πλαίσια ενός advisory forum, ενός συμβουλευτικού forum, το οποίο βοηθά το συντονισμό των καλύτερων εμπειρογνωμόνων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αξιολογήσεις επίσης αυτές κοινοποιόντουσαν, δημοσιεύονταν στην ιστοσελίδα του ECDC. Προσπαθούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουμε τι απαραίτητε συστάσει και την απαραίτητη καθοδήγηση στα κράτη-μέλη, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα των μελετών μα στι εθνικέ πολιτικέ ε, προστασία τη δημόσια υγεία. Επίση, πρέπει να σα πω ότι γίνανε πάρα πολλέ συναντήσει και συνεδριάσει. Δεν θέλω τώρα όμω να επιστέλθω σε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, Ακούσαμε πάρα πολλέ επικρίσει για του εμπειρογνώμονε, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα να περασπίσω όμω εμπειρογνώμονε, γιατί μα βοήθησαν πάρα πολύ, δείξαν έναν καταπληκτικό επαγγελματισμό και χωρί αυτού δεν θα είχαμε καταφέρει να καταλήξουμε στα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ε, Πρόσφατα είχαμε και το International Health Regulation, τους διεθνείς κανονισμούς για την ε, υγεία και την προστασία της δημόσιας υγείας, που θέτουν πλέον ένα διεθνές πλαίσιο για την κατάρτιση πολιτικών για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρέπει να σας πω ότι ε, η Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σαφώς είναι η πλέον αρμόδια για να κηρύξει το συναγερμό πανδημίας, αλλά καταλήγει στην απόφαση αυτή μόνο αφού συμβουλευτεί τους καλύτερους εμπειρογνώμονες. Και ακριβώς αυτό έκανε. Δεν λειτουργήσε κατά τρόπο αυτόνομο. Πρόεδρος, διακόπτη την ομιλήτρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Uh, Εάν talent. Ο κύριος Φλόρεντς, ναι, σε, τέτοιες, σε τέτοια διοικητικά θέματα είμαι ήρεμος, αλλά δεν ε, μπορώ να αποδεκτώ σήμερα το πρωί, ολόκληρο το πρωινό, κάποιοι συνάδελφοι να έχουν φέρει τηλεπτικές κάμερες και να μαγνητοσκοπούν τις ψηφοφορίες. Ε, ναι, εντάξει, είναι δημοκρατικό, αλλά να έρχεται μια κυρία και να κάθεται να βιντεοσκοπεί τον κατάλογο ε, συμμετοχών, πρέπει να σας πω ότι αυτό σε όλα τα χρόνια που συμμετέχω στο Κοινοβούλιο που το έχω ζήσει. Να ρωτήσουμε και να ρωτηθούμε ποιο κάνει κουμάντο εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο, θα είμαστε σύντομοι. Ποιο είναι λοιπόν υπέρ τη συνέχιση τη μαγνητοσκόπηση και τη φωτογράφηση. Ναι, δεν είναι θέμα, κύριε Λάιν. Το θέμα, καλοί φίλοι είμαστε, αλλά το θέμα δεν είναι να το αποδεχόμαστε. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες που μιλάνε για την ασυλία. Ναι, δεν χρειάζεται τεράστιες συζητήσει. Κοιτάω εδώ πέρα τι γίνεται, βλέπω τι γίνεται. Να παρακαλέσουμε την εν λόγω κυρία να βγει από την αίθουσα και να καταγραφή στα πρακτικά, λέει ο κύριος Φλόρεντς, ε, το όνομα της κυρίας αυτής. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Να περάσουμε λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε μάλλον για τις εισηγήσεις σας και να περάσουμε στον γύρο των ερωτήσεων. Θα είμαι αυστηρός και με τους βουλευτές όπως ήμουν αυστηρός και με τους προσκεκλημένους μας. Ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση και 30 δευτερόλεπτα επερώτηση και ένα λεπτό δεύτερη απάντηση. Η πρώτη ομιλήτρια. Αν γίνεται συγκεκριμένα σε κάποιον να θέλετε τα ερωτήματά σας. Μισελ, ένα λεπτό έχεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι ιδιαίτερα που γίνεται αυτή η ακρόαση. Η βασική ερώτηση που θέτω είναι η εξής. Είναι εξαρτώμενη ή ανεξάρτητη η Ευρώπη από τους διεθνείς οργανισμούς. Γιατί το πρόβλημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Η, Παγκόσμιο, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στις 11 Ιουνίου κήρυξε την πανδημία. 164 νεκροί 144 νεκροί συγγνώμη, σε 166 χώρες. Και βγαίνει λοιπόν εδώ συναγερμός επίπεδου 6 για πανδημία. Και εγώ λέω, ορίστε, ως βουλευτής, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά όργανα, η ΕΠΑ, το ΣΕΝΤΕΣΕ, η ΑΣΟΕΦ, η ΑΣΔΕΣΕ. Ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν, ποιος έχει την εξουσία για να πει συμφωνούμε με τον συναγερμό επίπεδου 6 για την ε, μαζική ή στοχευμένη ε, εμβολιασμό. Λοιπόν, ποιος είναι ο υπεύθυνο, ποιος θα απαντήσει, η Κομισιόν. Είναι καλό το ερώτημα, αλλά δεν είναι εύκολο να απαντήσω. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος ως Ευρωπαϊκή Ένωση της ΠΟΗ, αλλά όλα τα κράτη-μέλη είναι μέλη της ΠΟΗ. και οι σχετικέ συμβάσει έχουν υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη σχετικά με το συντονισμό τη αντίδραση στην κρίση αυτή. Και φυσικά, επειδή ήταν παγκόσμια η φύση της απειλής αυτής, είναι δύσκολο να πούμε ότι δεν ήταν κανεί υπεύθυνο για το συντονισμό. Η ΥΠΟ είναι η κατάλληλη ε, υπηρεσία για να λάβει αποφάσεις και αυτό συνέβη. η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της ακολούθησε το σχέδιο τιμότητας που εξήγησε ο κύριος Τζον Ράιαν, το οποίο είχε συμφωνηθεί το 2005, το οποίο αποτελούσε και τμήμα της ε, ανταπόκρισής μας στις διεθνείς συμβάσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν, θεωρώ, να διασφαλίσουμε ότι οι υπόλοιποι διαδραματίζει όσο καλύτερα γίνεται το ρόλο τη για να αντιδρούμε σε αυτές τις κρίσεις. Επερώτηση. Το συμπέρασμα που ανασύρω από την απάντησή σας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα εξαρτάται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Δεν έχει καμία εξουσία να πει διαφωνούμε με αυτό το οποίο αποφασίσατε. Ε, λοιπόν, γιατί πληρώνουμε τα ευρωπαϊκά όργανα η ε, κυρία Λάλιν, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε ιδιαίτερα, αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε όλο τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλοί εμπριογνώμονες στη δημόσια υγεία, στα κράτη-μέλη. Και δεν υπήρξε αμφισβήτηση της ε, σχετικής μελέτης που είχε κάνει Αυτό το υπογραμμίζουμε. Ευχαριστώ κυρία Γιάκοπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω εκ νέου το εξή. Η αξιολόγηση κινδύνου στα πλαίσια του ECDC ήταν ανεξάρτητη, αλλά εξετάσαμε τα ίδια δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους και όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί. Άρα καταλήξαμε σε παρόμοια πορίσματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν κάναμε ανεξάρτητη αξιολόγηση κινδύνου. Δεύτερο στοιχείο που ήθελα να τονίσω. Η ΠΟΗ συνήθως ε, λειτουργεί με ομοφωνία. Δεν υπάρχουν πολλά δεσμευτικά εργαλεία στην ΠΟΗ. υπάρχει, υπάρχουν κάποια στα οποία συμμετέχουν και τα κρατημέλη και φυσικά υπάρχει σχετική ευελιξία. Να τονίσω λοιπόν ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε λεπτομερώς αυτό το σύστημα ευελιξίας για την επόμενη ευελιξία, την επόμενη κρίση. Η... Στο νότιο ημισφαίριο συνεχίζεται ακόμα η κρίση, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προετοιμάσουμε την τοπική διάσταση αυτού του παγκοσμίου πλαισίου για την επόμενη κρίση. Αυτό πραγματικά είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εργαστούμε πιο εντατικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελβό, σκιώδης από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι κάπως ε, πιο σκεπτική στρία για τη συνεργασία των κρατών μελών και θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας που αποτελεί ένα όργανο κλειδί για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών μια για τη συνοχή στη δουλειά τους. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή έχει την καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα. Ε, Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ομόφωνα σε αυτήν την Επιτροπή έγιναν σεβαστές ε, στα κράτη-μέλη. Μετά ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη μετά από την απόφαση ο καθένας στη γωνιά του πήγε και να, κατασκευάσει το δικό του, να παρασκευάσει το δικό του εμβόλιο. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ε, θα αρκεί το στόκ το οποίο έχουμε. Ποιος θα απαντήσει? Η κυρία Τέστο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ζητώ συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι προχωράμε τώρα αυτή τη στιγμή στο ζήτημα του επόμενου πάνελ. Δύο πράγματα μπορώ να πω πάντως. Βάσει των νέων άρθρων της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει να κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου προκειμένου να εγκρίνει μέτρα για να αντιμετωπίσει μια δυσυνοριακή πανδημία. Επομένω, εμεί, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνουμε μια πρόταση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο βάσει του νέου αυτού άρθρου τη συνθήκη τη Λισαβόνα, προκειμένου να έχουμε έναν κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν την πρόταση αυτή και θα την παρουσιάσουμε του χρόνου, γιατί είναι πολύ πολύπλοκη. Αν είχαμε λοιπόν το άρθρο αυτό και τον κανονισμό, θα είχαμε αποφασίσει εμείς για τη δική μας την αντίδραση, ακόμα και αν ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είχε άλλη στάση. Θα μπορούσαμε να είχαμε δηλαδή μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή κοινωνική, ε, συγγνώμη, κοινοτική αντίδραση και τοποθέτηση. Δεν μπορούσαμε όμω να κάνουμε κάτι τέτοιο, κάτι εντελώ ανεξάρτητο και δεν υπήρχε νομική βάση. Για το εμβόλιο θα μιλήσω στην επόμενη παρέμβασή μου. Reaction. Άρα το εγώ αυτό το πράγμα είναι ότι πρέπει να δακτυλοδείξουμε το τι δεν ε, λειτουργήσε μέχρι τώρα για να το διορθώσουμε σε μία επόμενη δράση. Μια άλλη ερώτηση τώρα, σχετικά με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η οποία μέσα από συγκεκριμένο ορισμό της πανδημίας όρισε το επίπεδο της, ε, ε, του συναγερμού. Όχι λόγω των αποτελεσμάτων που είχε μέχρι τότε, αλλά ε, με κριτήριο την ταχύτητα ε, διάδοσης, γιατί κανένας δεν μπορεί να προβλέψει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ερώτηση, όχι, για διαπίστωση είναι. Κυρία Γιάκοπ. Να σας πω ότι ε, τα κριτήρια για μια πανδημία είναι τρία. Πρώτον, πρέπει να έχουμε έναν ιό. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και τρίτον, να έχουμε και την γεωγραφική διάσταση. Όλα αυτά τα βλέπουμε στις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Κανονισμού για την Αντιμετώπιση των Κρίσεων στη Δημόσια Υγεία. Τον Ιανουάριο και τον Μάιο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βασίστηκε στα κριτήρια αυτά και ήμασταν σε θέση κατά αυτόν τον τρόπο να εμπλουτίσουμε περισσότερο τις, α, τους διεθνείς κανονισμούς για την υγεία. Αυτά είναι πάντως τα κριτήρια και θα μπορούσαμε όμως να τα εμπλουτίσουμε με άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα η σοβαρότητα της νόσησης. Κάτι στο οποίο θα ήθελα να αφαιρθώ κύριε Πρόεδρε, είναι ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές αποφάσεις στα εθνικά μέτρα των κρατών μελών. Και αυτό γιατί από τη μία χώρα στην άλλη η ποσότητα των εμβολίων διέφερε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη είχαν διαφορετικές προτεραιότητες. Βάσει του αριθμού των εμβολίων που είχαν έπρεπε να αποφασίσουν ποιον θα εμβολιάσουν κατά προτεραιότητα. Και αν δούμε τι γίνεται σε όμορες χώρες είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες για ποιο λόγο σε μια γειτονική τους χώρα αποφάσεις είναι τελώς διαφορετικές. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερη συνέργεια, καλύτερο συντονισμό των υγειονομικών μέτρων από τη μία χώρα στην άλλη και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα επικοινωνίας. Θεωρώ ότι η επικοινωνία δεν ήταν καλή. Ισκιώδης από τους σοσιαλιστές, η κυρία Κάντα. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τους εκπροσώπους των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήθελα να πω, η κυρία Κάντμπαχ, ότι σήμερα κοιτάμε πόσα εκατομμύρια εμβόλια δεν χρησιμοποιήσαμε στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, αλλά κοιτώντας τι λέγεται σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. γιατί σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί η άποψη ότι δεν υπήρχε λόγος για την ιστερία αυτή που προκλήθηκε. Ρωτώ λοιπόν, για να περάσουμε ίσως και λίγο προς το δεύτερο τμήμα, η <coughs> ευρωπαϊκή θεσμοί είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αυτή την εξωτερική διάσταση, το πώς έγινε αντιληπτή η κρίση και κατά δεύτερον χρειαζόμαστε μήπως επιπλέον αρμοδιότητες για να είναι πιο ρεαλιστική αυτή η εικόνα που δώσαμε προς τα έξω και πώς θέλουμε, πώς ε, σκοπεύουμε να ξαναβρούμε την αξιοπιστία που χάσαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Πρόεδρος. Περνάμε λοιπόν λίγο και στον επόμενο γύρο που αφορά το μέλλον. Ποιος θέλει να απαντήσει, κύριε Ράιεν. Yes. Σε ό,τι αφορά το τμήμα που αφορά το παρελθόν. Απάντηση. Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τις ε, ασθένειες της μολυντικής. ασθένειες βασίζεται και επηρεάζεται και από την στρατηγική της Λισαβόνας, την συνθήκη της Λισαβόνας. Κοιτώντας λοιπόν τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε με την συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να ενισχύσουμε την νομοθεσία για να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει σε τέτοιες καταστάσεις. Η κυρία Γιάκοπ να πω εν συντομία ότι και εμείς είχαμε πολλές αβεβαιότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Να το έχουμε αυτό υπόψη. Είχαμε λίγες πληροφορίες για το πώς θα διαδίδονταν η, η πανδημία και πόσο επικίνδυνη θα ήταν. Όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη. Ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα σενάριο πολύ χειρότερο από αυτό που τελικά διαμορφώθηκε. Ωστόσο, είχαμε την υποχρέωση να εφαρμόσουμε την αρχή της πρόληψης για να προστατεύσουμε τις ζωές των πολιτών. Και αυτή ήταν η λύση που επέλεξαν όλοι οι θεσμοί. Ωστόσο το βασικό μου μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στο μέλλον για να διασφαλίσουμε ότι αν υπάρχει πιο ήπια κρίση Εμεί θα είμαστε προετοιμασμένοι πολύ παραπάνω για να είμαστε σε θέση να δράσουμε. Σωστά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλη επερώτηση, λέει ο Πρόεδρο, και να περάσουμε στην Κορίν Λεπάζο από του Φιλελεύθερου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι για αυτήν τη δημόσια κρόαση. Ρωτώ την κυρία Γιακόμπ. Κυρία Διευθύντα, Εγώ διάβασα προσεκτικά το λόγο σας και τις απαντήσεις που δώσατε και ήσασταν ιδιαίτερα μέτριοπαθείς για την εξέλιξη και τα πραγματικά ρίσκα για πανδημία της γρήπης. Γιατί αυτή η μετριοπαθής λοιπόν άποψη δεν είχε μεγαλύτερες επιπτώσεις. Δεύτερον, ήσασταν ιδιαίτερα ακριβείς ε, στα ρίσκα που έχουν να κάνουν με τις παρενέργειες και και ποιο, ποιοι έπρεπε να εμβολιαστούν. Και λέγατε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τους υγιείς ενήλικες. Γιατί δεν ελήφθη υπόψη αυτή η θέση. Και μία ασάφεια, ασυμβατότητα συγγνώμη, που με ενοχλεί. Λοιπόν, περνάτε εσείς από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 2 και μετά ξανααλλάζετε μετά από μερικούς μήνες. Και μετά, μέσα σε μερικές μέρες εσείς αναγγέλλετε ότι θα ακολουθήσετε την OMC, ε, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να περάσετε σε επίπεδο 6. Το γεγονός ότι αυτά τα οποία δηλώσατε δεν είχαν συνέχεια ή είναι μια συνειδητή επιλογή και, και τι... Κυρία Γιάκομπ. Ο ρόλος του ECDC για την ε, αξιολόγηση κινδύνου ε, δεν, ε, μάλλον αυτό που λέτε δεν εντάσσεται στην παιδιαρμόδιότητα του ECDC, γιατί είναι σύμφωνο το περιβάλλον Υπάρχουν υπηρεσίε όπω είναι το ACDC που αξιολογούν του κινδύνου και παρέχουν επιστημονικά στοιχεία και συστάσεις, αλλά στη συνέχεια τα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνα για την διαχείριση κινδύνου και για τι αποφάσει ε, δημόσια υγεία λαμβάνουν τελικά τι αποφάσει με το συντονισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επειδή τα κράτη-μέλη όλα εντάσσονται και συμμετέχουν στην σχετική νομοθεσία για την δημόσια υγεία, τη διεθνή, από κοινού αποφάσισαν να περάσουν στη φάση 6 και θεωρώ, όπως είπα και προηγουμένως, ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ περισσότερη ευελιξία στα εθνικά σχέδια εθνικής ετοιμότητας για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και εθνική αλλά και τοπική ε, ευελιξία και το διεθνές πλαίσιο προβλέπει τέτοιες δυνατότητες. Αν δούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο σωστό να περάσουμε από την φάση 5 στη φάση 6, Μπορεί να γίνει αυτό και να το κάνουμε αυτό σε ό,τι αφορά τα σχέδια εθνικής ετοιμότητας. Να τα σκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά και να σκεφτούμε και με τους υπόλοιπους φορείς πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα, αλλά υπάρχουν πιο πολλά σε ό,τι αφορά την... Μάλλον δεν είναι μόνο η εξελόγηση κινδύνου, στην διαχείριση του κινδύνου. Ευχαριστώ για την απάντησή σας, αλλά συγγνώμη, δεν είναι απάντηση λέτε δεν είναι ευθύνη του ΣΕΝΤΕΣΕ, το καταλαβαίνω, εντάξει. Αλλά γιατί, τι έγινε, τι μεσολάβησε σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε αυτά τα οποία είπατε δεν ελήφθησαν υπόψη. Ποιος μπλοκάρισε όλα αυτά. Θέλουμε να ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι κόλλησε πουθενά το θέμα, γιατί οι πληροφορίες αυτές ήταν πάντα γνωστές στα κράτη-μέλη. Και όλα αυτά ήταν γνωστά στο ευρωπαϊκό σύστημα. Κάθε μέρα γίνονταν βιντεοδιασκέψει κατά τη διάρκεια τη κρίση με τα κρατημέλη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε μέρα αναθεωρούσαμε την κατάσταση και τα μέλη του συστήματος έγκυρης αντιμετώπιση που λαμβάνουν τι αποφάσει τα κρατημέλη καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι και συζητούσαν τις απαραίτητες δράσεις, τα απαραίτητα μέτρα. Οι συμβουλές ε, του ECDC ήταν τεχνικής φύσεως. Αυτό είναι ο κανόνας που μας διέπει. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το σύστημα δούλεψε. Ναι, να δώσουμε το λόγο στη Σουηδική Προεδρία, λέει ο Πρόεδρος. Thank Σας ευχαριστώ. Όπως υπόθηκε ήδη, η διαχείριση του κινδύνου γίνεται κυρίως από τα κράτη-μέλη, είναι αρμοδιότητα κυρίως των κρατών μελών. Δεν υπάρχει όμως κάποια βασική διαφωνία ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες ότι έγινε κακή αξιολόγηση από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όλοι οι παγκόσμιοι εμπειρογνώμονες συμφωνούσαν ότι όντως μιλούσαμε εκείνη την εποχή για απειλή και τα κράτη-μέλη αντέδρασαν αναλόγως και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε την αντίδραση ενός ιού. Ενδεχομένως και την επόμενη φορά να έχουμε ακριβώς την διαβεβαιότητα, ακόμα και να έχουμε ευέλικτα σχέδια. Και σαφώ θα πρέπει να αποκομίσουμε τα σωστά διδάγματα. Και σαφώ θα πρέπει στα κριτήρια να συμπεριλάβουμε και τη σοβαρότητα. Καταλαβαίνετε όμω ότι πάντα θα υπάρχει ένα βαθμός αβεβαιότητας και σε ένα κλίμα βεβαιότητας θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσει και ακριβώ αυτό κάναμε ήταν μια υπεύθυνη απόφαση που ελήφθη στα πλαίσια των συγκεκριμένων συνθήκων αβεβαιότητας. Ευχαριστούμε. Ο τελευταίος ε, σκιώδης είναι η Μαρίζα Ματίας από την ΚΟΕ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να συγχαρώ για την οργάνωση αυτής της ακρόασης. Εγώ πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε για το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όλη αυτή τη διαδικασία υπέσκαψε την αξιοπιστία τους. Φτάνει να δει κανείς ποια ήταν η αντίδραση του κοινού μετά από τα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν για την Παρασκευή των εμβολίων. Και ποιο ήταν δηλαδή το αποτέλεσμα μετά. Εξήγησαν όλοι ποια μέτρα ελήφθησαν, τι κάνανε προσπάθησαν να διαχειριστούν μια κατάσταση αβεβαιότητας αλλά επτόχευσαν ε, στην διαφάνεια. Αν, υπήρξε, αν υπήρχε πραγματική διαφάνεια και πληροφόρηση, δεν θα χρειαζόταν καν να έχουμε αυτή την ακρόαση. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ αποτελεί την απόδειξη της πτώχευσης όλης αυτής της πολιτικής. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν σήμερα για να ανακτήσουμε την εμπειρία των πολιτών η οποία χάθη πλήρως. Um Υπάρχει συνταγή για να ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία άραγε. Έχει τεθεί το ερώτημα λοιπόν και θα το απαντήσει με το ερώτημα όταν θα μιλήσουμε για το μέλλον. Δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο για να την απαντήσει πάρα αυτά. Εύκολα χάνεται η αξιοπιστία, αλλά δύσκολα ξανακερδίζεται. Το ξέρουμε αυτό και στην πολιτική μία επιπλέον παρατηρήση. Η Μαρίζα είχε μισό λεπτό παραπάνω. Δεν με ακούει όμως. Εντάξει, να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Τα μαθήματα που θα πρέπει να αντλήσουμε για το μέλλον. Θέλετε να δευτερολογήσετε, Μαρίζα. Μα εμένα δεν μου απάντησε ακόμα κανεί την ερώτησή μου και να κάνω και μία επερώτηση αν συμφωνείτε. Γιατί όχι μόνο δεν έχουμε πληροφορίες και διαφάνεια, αλλά και οι ερωτήσεις που έγιναν πριν δεν απαντιούνται. Ρωτώ το μοντέλο παρέμβασης μπορεί να χρησιμοποιείται σε αντίστοιχες καταστάσεις και τι γίνεται μετά και με τις ερωτήσεις οι οποίες ε, δεν απαντήθηκαν από το πάνελ. Κύριε Ρίς, θέλει να τολμήσει να δώσει απάντηση. Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω την ερώτηση αυτή καλύτερα είναι να ακούσουμε και τον επόμενο γύρο, αλλά να επανέλθω στο παρελθόν. Το πιο δύσκολο τμήμα ήταν η επικοινωνία με το κοινό και με τους ε, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Όταν ξεκίνησε στις αρχές του Ιουλίου το Βαλγικό, η Βελγική Σύνοδος, ήταν δύσκολο να βρεθεί ακόμα και ορισμός και όνομα για τον ιό. Γιατί στην αρχή το ονομάζαμε η, ο ιός των ε, χείρων. Η γρήπη των χείρων. Μετά στη συνέχεια ονομάστηκε Μεξικανική γρήπη. Μετά ή τα ένα 1 ένα. Και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικός ορισμός στις διάφορες γλώσσες. Στα αγγλικά και στο διαδίκτυο επικρατούσε όρος swine flu, η γρήπη των χείρων. Οι διάφορες ομάδες και οι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας δεν ήταν επαρκώς πληροφορημένοι. Δεν είχαν πρόσβαση στις πληροφορίες ή ίσως να μην είχαν έγκαιρη πρόσβαση ή ίσως να μην είχαν χρόνο να αφιερώσουν στην πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Και αυτό ήταν ένα σημείο κριτική σε όλες τις χώρες, σε πολλές τις χώρες. Ένα τρίτο φαινόμενο στην πανδημία αυτή ήταν τα κοινωνικά μέσα. Το Facebook είχε ήδη συμμετάσχει. Πολύ απευθύνοντας το κοινό ως εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και να περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο σχετικά με τα μαθήματα που αντλήσαμε. Βασική ερώτηση είναι ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην σχεδιασμό αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία, την αριστεία και την διαφάνεια της διαδικασίας λήψεων αποφάσεων. Η κυρία Πάολα Πεστόρη, θα πάρει το λόγο. Τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη σημερινή συζήτηση το πιο σημαντικό είναι να δούμε ότι όντω στο παρελθόν έχουμε επικρίσει, ακούσαμε όμω και συγχαρητήρια, θα πρέπει να τανίσουμε και το μέλλον. Για το μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει κάποιε πρωτοβουλίε οι οποίε δείχνουν ότι έχουμε αντλήσει πλέον διδάγματα και ότι είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την απόκρισή μα. Πρώτον, από γενική απόψεω έχουμε πλέον ένα άρθρο συνθήκη Λισαβόνα και επομένω μια νέα αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποβάλουμε μια μονοθετική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει καλύτερο στονισμό και καλύτερη ανταπόκριση σε κοινοτικό επίπεδο. Επίση, θα ήθελα να σα επενθυμίσω ότι ε, η Health Security Committee, η Επιτροπή Ασφάλεια Υγεία, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Ντελβό, αυτή τη στιγμή εργάζεται βάσει συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Δεν έχει επίσημο νομικό καθεστώ. Εργάζεται η Επιτροπή αυτή, λειτουργεί καλά ω μηχανισμό, αλλά η νομική, η τη βάση είναι πάρα πολύ ασθενή ακόμα γιατί βασίζεται απλώς σε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Στο νέο νομοθετικό πακέτο που θα προτείνουμε του χρόνου, θα προτείνουμε και μια νομική βάση για την Επιτροπή αυτή για να υπάρχει καλύτερο τονισμός με τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, πρέπει να εργαστούμε περισσότερο στον τομέα των εμβολίων. Είδαμε στο παρελθόν ότι τα κράτη-μέλη βρισκόντουσαν σε μία άδικη θα έλεγα κατάσταση όσον αφορά τις συμφωνίες αγοράς, όσον αφορά τις ρήτρε επιστευτικότητας που έπρεπε να υπογράφουν. Δεν υπήρχε αρκετή διαφάνεια όσον αφορά την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Επομένως εμείς επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή έναν κοινό μηχανισμό προμήθειας εμβολίων που θα μπορούσε να συμπεριλάβει και ένα σύστημα επαφής μεταξύ κρατών μελών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ένα στόκ, ένα απόθεμα σε κοινοτικό επίπεδο, το οποίο θα μπορούσε να διοικητευτεί στις χώρες που το έχουν ανάγκη. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Τρίτον, το ζήτημα του σχεδιασμού της ετοιμότητας. Ο σχεδιασμός ετοιμότητας υφίσταται προφανώς σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και εδώ πάλι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών είναι οι πιο σημαντικές. Έχουμε ένα κοινό σχέδιο, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πίσω ότι υπάρχει και μια ισχυρή νομική βάση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό. Ένα σημείο τώρα που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το συντονισμό ήταν οι στρατηγικές εμβολιασμού. Σε σχέση με αυτές, τα κράτη-μέλη στο παρελθόν είχαν το καθένα μια ξεχωριστή στρατηγική. Σαφώς υπήρχε ανταλλαγή ε, πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και πάλι λυπάμαι θα σας το πω, δεν υπήρχε η κατάλληλη νομική βάση προκειμένου να πετύχουμε τον κατάλληλο συντονισμό. Πολλές φορές αυτή η νομική βάση δεν υφίστατο καθόλου. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε εδώ ένα μηχανισμό πολύ πιο ισχυρό. Και τέλος, η ανακοίνωση προς τα έξω, προς το κοινό, πληροφορίες προς το ευρύτερο κοινό. Δεν λειτουργήσε καλά το σύστημα αυτό, δεν ήμασταν σε θέση να δώσουμε το σωστό μήνυμα προς τον Ευρωπαίο πολίτη, όχι μόνο προς το κοινό, ακόμα και στους ίδιους τους επαγγελματίες της υγείας, γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη επαγγελματίες της υγείας λάβανε διαφορετικές αποφάσεις. Θα έχουμε λοιπόν μια νέα νομική βάση, βασιζόμαστε πλέον σε ένα νέο άρθρο της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα έχουμε ένα κοινό σχέδιο προμήθειας εμβολίων και ένα καλύτερο επικοινωνιακό σχέδιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Τεστόρη. Σαφώς τα κράτη-μέλη έχουν μια πολύ σημαντική ευθύνη, ο κύριος Ράινερς εξ ονόματος Βελγικής Προεδρίας. Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ε, εκφράσω τη συγγνώμη της κυρίας Όνκε η οποία είχε προγραμματίσει να έρθει, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να έρθει. Να συμμετέχει δηλαδή σε αυτήν την τόσο σημαντική συζήτηση. Όπως ξέρετε πολύ καλά η Βελγική Προεδρία στις 2 Ιουλίου μαζί με την Κομισιόν οργάνωσε μια τεχνική ε, διεθνή διάσκεψη για αυτό το θέμα και είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν μέλη της Επιτροπής σας. Πάνω από 300 εμπειρογνώμονες από τρίτες ε, χώρες, διεθνείς οργανώσεις κλπ. ήταν παρόντες. Και όλοι ε, κλήθηκαν να ανασύρουν το συμπέρασμα της ε, πανδημίας ε, του 2009 και να εμπλουτίσουν με τα συμπεράσματά τους ε, τη συζήτηση του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου τα στείλαμε στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η οποία ασχολείται με την εξέταση ε, του διεθνούς ε, κανονισμού για τις ε, πανδημίες υπό το φως δηλαδή αυτής της πανδημίας. Να σας πω τώρα ποια ήταν τα συμπεράσματα των Υπουργών. Καταρχήν θέλω να υπογραμμίσω ότι η αποτελεσματικότητα των εθνικών πολιτικών για την πανδημία γρήπης αμφισβητήθηκαν από τις πολιτικές των γειτονικών χωρών. Ο συντονισμός, όπως το ξέρετε, δεν ήταν ε, το, το, το, γερό σημείο όλης αυτής της ιστορίας. Και επίσης υπήρξε ένα πρόβλημα συνεργασίας με τους διεθνούς οργανισμούς, με τους διεθνούς οργανισμούς και λοιπά. Διότι όταν μιλάμε για πανδημία δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά. Η πανδημία είναι κάτι το οποίο εξαπλώνεται με φοβερή ταχύτητα, άρα πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια. Λοιπόν, μερικά από τα διδάγματα χρειάζεται. παρακολούθηση, προ, ε, προληπτική παρακολούθηση για να λαμβάνετε υπόψη η πανδημία στην πραγματική της διάσταση. Επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και του υπολείπου κόσμου σε όλα τα επίπεδα για τις ε, πληροφορίες, ε, σε όλα τα υγειονομικά επίπεδα. Τώρα, ε, η... πρέπει να ενισχυθεί η επικοινωνία, πρέπει να η χρήση των εμβολίων συζητήθηκε πάρα πολύ στα κράτη-μέλη και πρόκειται για έναν τομέα όπου η συνοχή και η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα. Στόχος ε, του μηχανισμού κοινών αγορών που είχε αποφασίσει το Συμβούλιο και τον έφερε η κυρία Τεστόρη <coughs> δεν διασφαλίζει μόνο μια μεγάλη συνοχή αλλά ενισχύει και την ποιότητα των εμβολίων. Τα κράτη-μέλη υπό την πρόθεση της Βελγικής Προεδρίας δέχθηκαν να συνεργαστούν με την Κομισιόν και τους οργανισμούς της για μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε περίοδο κρίσης. Διαφάνεια στην πληροφόρηση αποτελεί πρόκληση για το μέλλον. Το λέει αυτό και το, ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν δεσμεύθηκαν. Ευχαριστώ, διακόπτει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λονγκρίν από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ. Η Βελγική Προεδρία τόνισε την ανάγκη να συμμετέχουν οι πρόσωποι των ε, ασθενών και οι επαγγελματίε στον τομέα της υγείας. Το εξετάζουμε αυτό ενεργά και θέλουμε περισσότερα. Μια άλλη σύσταση ήταν να οριστεί καλύτερα ο ρόλος των εθνικών αρχών του SDC και ο το και εγώ εργαζόμαστε στενά για να εξετάσουμε πώς μπορούμε να ε, εναρμονίσουμε τις ε, αντιδράσεις μας προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα σε μελλοντική πανδημία για να κοιτάξουμε σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Θα χρειαστούμε πιο μεγάλη ευελιξία. Η στρατηγική έχει καταρτιστεί για το χειρότερο σενάριο και η πρόσφατη εμπειρία μας καταδεικνύει ότι πάντα θα επικρατεί ε, αβεβαιότητα για, την, για τους ιούς της πανδημίας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για διαφορετικά στελέχη της γρήπης και θα πρέπει να υπάρχουν σωστές κλινικές μελέτες προτού ξεσπάσει νέα πανδημία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους σχετικούς εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι σαφές ότι η σχέση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό και τη σχετική στρατηγική. Και γι' αυτό θα είναι σημαντική και η επικοινωνία με το κοινό. Θα πρέπει να ενισχυθεί. Κοίτοντας το μέλλον, σκοπός είναι όλοι οι μηχανισμοί να επιταχύνουν την ε, διαθεσιμότητα των εμβολιασμών και θα πρέπει επίσης να δετίθενται ε, καλύτερα στοιχεία από τις κλινικές μελέτες. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το κλινικό πρωτόκολλο για την δοκιμή των εμβολίων και επίσης σε ό,τι αφορά την έγκριση. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα συστήματα αναφοράς ε, προβλημάτων και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία αυτή. Και θα πρέπει να βελτιώσουμε τις μελέτες μας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την βιομηχανία προς τον τομέα της μελέτης. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες και συντονισμένες μελέτες για να εξασφαλιστεί ότι θα ενημερώνονται διαρκώς οι πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα. Τέλος, θα πρέπει να διατίθενται τα κατάλληλα στοιχεία για την ασφάλεια των εμβολιασμών σε ό,τι αφορά την ανοσοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα περνάμε στο νέο επικεφαλής του ECDC, τον κύριο Σπρέγγερ, για τις μελλοντικές δράσεις του ECDC. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Τρία διδάγματα εγώ μπορώ να δω για το ECDC. Πρώτον, οι εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας θα πρέπει να κάνουν πιο πολύπλοκες αξιολογήσεις του κινδύνου πολύ πιο νωρίς πριν την εκδήλωσή του. Και θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό λίγο αργότερα όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου. Δεύτερο μάθημα. Η δική μας ανάλυση του επίπεδου του κινδύνου που δικαιολογεί τις δημόσιες δαπάνες και την εκστρατεία εμβολιασμού για το σύνολο του πληθυσμού ή για συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο πιο πολύπλοκο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα να γίνεται μια κοινωνικο-οικονομική ανάλυση για τις εκστρατείες εμβολιασμού. Σε περίπτωση πανδημίας ή σε οποιαδήποτε άλλη έκτακτη κατάσταση εμβολιασμού είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται επίσημοι έλεγχοι για το αν έχει γίνει κάποια αναθεώρηση αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο παρελθόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν κάποιες νέες πληροφορίες, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναθεωρούμε και να επικαιροποιούμε τις αποφάσεις που έχουμε λάβει στο παρελθόν. Και τρίτον, η πολιτική επικοινωνία που έχουμε θα πρέπει και αυτή να αναθεωρηθεί. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε καλύτερα ποια μηνύματα περνάνε προς τους ανθρώπους και ποια μέσα χρησιμοποιούνται περισσότερο. Επίσης η πανδημία μας δίδαξε ότι και οι ίδιοι επαγγελματίε της υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες. Αν δεν να πιστούν από τα μηνύματα που στέλνουμε εμείς, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πιστούν οι ασθενείς. Πιστεύω πάρα πολύ στα συστήματα επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο. Πρώτο λοιπόν δίδαγμα, πρέπει να γίνεται πολύ νωρίς μια πολύ καλύτερη ανάλυση του κινδύνου για την επόμενη πανδημία γρήπης, το ECDC προτίθεται να χρησιμοποιήσει περισσότερες παραμέτρους στην αξιολόγηση του κινδύνου και όχι μόνο δεν θα κάνει απλώς μία αξιολόγηση των κρουσμάτων και της γεωγραφικής επέκτασης ε, του ιού. Αυτή η πιο πολύπλοκη, η καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου προποθέτει ότι θα χρησιμοποιούνται περισσότεροι παράγοντε και περισσότερα κριτήρια στην αξιολόγηση του κινδύνου και σαφώ το ECDC θέλει να συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση του συστήματο αξιολόγηση. Μπορείτε επίση να δείτε και το μελλοντικό πρόγραμμα του ECDC όπου προβλέπεται συγκεκριμένο προπολογισμό για την καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου στο μέλλον. Επίση θα ήθελα να σα πω ότι οι εθνικοί οργανισμοί υγεία και τα εργαστήρια τα οποία συνεργάζονται κάθε φορά είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντε. Μόνο μέσω αυτών των εθνικών κέντρων δημόσιας υγείας και μόνο μέσω των εθνικών εργαστηρίων θα καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη ετοιμότητα. Βασίζεται σε αυτά τα δεδομένα και το ECDC προκειμένου να κάνει καλές αξιολογήσεις. Πιστεύω ακόμα ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο βελτίωση στο μέλλον και νομίζω ότι η στάση μας θα πρέπει να είναι μετριοπαθής. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος, όντως έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα στο μέλλον. Ας επιστρέψουμε τώρα στις ερωτήσεις. Πρώτα η Σκιώδης, η κυρία Ντελβό πρώτα όσον αφορά τις μελλοντικές δραστηριότητες. Χαίρομαι για, τον, ε, για, για τις ε, ενισχυμένες ε, αρμοδιότητες στο μέλλον του οργανισμού. Χαίρομαι για το επίπεδο προβληματισμού στο Συμβούλιο, αλλά θέλω να πω το 2001 και το 2005 η Κομισιόν πρόθεσε τα κράτη-μέλη για έναν καλύτερο συντονισμό. Και πάλι το 2010 εδώ είμαστε και συζητάμε τα ίδια πράγματα και βλέπουμε να έχουμε τα ίδια κενά. Υπάρχει λοιπόν σήμερα μία πραγματική βούληση, διότι χωρίς αυτήν δεν θα προχωρήσουμε ποτέ. Εμείς διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν εντελώς αντιφατικές ε, ε, πληροφορίες και αποφάσεις για τον εμβολιασμό. Ε, υπήρξαν δυσκολίες λοιπόν και η πληροφόρηση είναι σημαντική, αλλά μπορούμε να έχουμε και ένα ενιαίο μήνυμα που μπορούμε να μεταδίδουμε, ένα ενιαίο μήνυμα το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται. Το πρόβλημα ήταν τελικά τι, η απώλεια εμπιστοσύνη του κοινού. Κυρία Τεστόρη. Ναι, Μιλώ εξ, ονόματο και τη Προεδρία, αν μου το επιτρέπει και ο κύριο Ράινε. Ναι, υπάρχει πολιτική βούληση και αυτό το καταδεικνύουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν πριν από δύο εβδομάδες μετά από την ανεπίσημη υπουργική συνάντηση του Ιουλίου υπό τη Βελγική Προεδρία. Ναι, και στην ανακοίνωση αυτού του Συμβουλίου ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει πρόταση για τις δημόσιες συμβάσεις. Ναι, είναι σωστό. Τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν να υπάρχουν τέτοια συστήματα, αλλά τώρα μας το ζητούν. Υπάρχει πολιτική βούληση. Χαίρομαι κάθε φορά που διαβάζω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου πάντα βρίσκω την ίδια, ε, την ίδια φράση. Ελπίζω λοιπόν να τα παρακολουθήσετε όλα αυτά από κοντά. Ο κύριος Ρέντερς. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε η κυρία Τεστόρη εξ ονόματος της Βελγικής Προεδρίας εγώ. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι δεν έχουμε φτάσει σε μία ενιαία θέση των 27 κρατών της Ένωσης για τη διαχείριση μίας κρίσης. Αυτό είναι φανερό. Αλλά <coughs> πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες του 2001 και το 2005 βοήθησαν να προχωρήσουμε τα πράγματα. Δεν είμαστε πια 27 διασκορπισμένοι έχουν γίνει προσπάθειες, ο κύριος ο Δόκτωρ Ράιαν τα παρουσίασε στην εισαγωγή. Υπάρχουν κάποιες ανεπάρκειες. Τα γεγονότα όμως που ζήσαμε πέρυσι μας ε, προωθούν να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε να καλωσορίσω τους ε, προσκεκλημένους μας. Αυτό που ακούμε είναι ωραία στη συζήτηση, αλλά ποιος θα έλεγε πέρσι κατά τη διάρκεια της ε, πανδημίας ότι α, να κάτσουμε λίγο και να μην υπερβάλλουμε και να μην κάνουμε τίποτα. Και για να είμαστε ειλικρινείς ότι η ΠΟΗ δεν αποτελεί για μας αρχή, αλλά ούτε αυτό είναι καινούργιο για μας. Χρειάζεται μια υπηρεσία που θα καλύψει τις ανάγκες όλες της Ασίας, όλης της Αφρική, Αφρικής και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να μας αρκέσει αυτό. Όχι. Όχι, αυτό το γνωρίζουμε. Δεν είναι καινούριο. Η αίμα θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί όταν θα χρειαστεί. Και αυτό είναι αποδεκτό. Και για το ECDC έχει δίκιο ο κύριος Φρέγκερ όταν λέει ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου. Αλλά τα βασικά στοιχεία τα είπαν ο κύριος Ράινερ και η κυρία Τεστόρη. Αν δεν υπάρχει νομική βάση, αν τα κρατημέλη δεν θέλουν να συνεργαστούν, δεν θα προχωρήσουμε καθόλου. Αυτό είναι το απλό μήνυμα. Τα υπόλοιπα είναι και ένα λόγια. Χρειαζόμαστε νομική βάση, χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία και πρέπει να δηλώσουμε πού βρισκόμαστε. Και ότι βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε λόγω των κρατών μελών. Τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Είναι αυτονόητο αυτό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια απάντηση ή κάποιο σχόλιο. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να απαντήσει, Πρόεδρε. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικά σαφές ε, το περιεχόμενο της συζήτησής σας. Κύριε Λεπάζου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσυπογράφω απόλυτα αυτό το οποίο είπε η Ντάγμαχ. Αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο μας είπε ο Διευθυντής της ΕΝΤΕΣΕ. Διότι όλα εντάξει μια χαρά, αλλά ό,τι κάναμε μέχρι τώρα στήχησε του σε όλη την Ευρώπη. για να είμαστε δηλαδή αποτελεσματικοί για την αντιμετώπιση των, ανεσ... ασθενειών. Εγώ κύριε Διευθυντά θέλω να σας ρωτήσω, μα τι σας χρειάζεται για να μπορείτε να είστε απόλυτα λειτουργικό σε αυτό το επίπεδο και να έχετε και μία ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη γνωστή από το ευρύ κοινό. Εμείς χρειαζόμαστε βεβαιότητα για την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων και των κατασκευαστών των εμβολίων. Δεν μιλήσαμε εμείς για την ευθύνη, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν το εξετάσαμε καθόλου. Θέλουμε λοιπόν ανεξαρτησία και καλή διάδοση και ενημέρωση του κοινού. Ποιος θέλει να απαντήσει, ο κύριος Σπρίγκερ. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στο ECDC είναι ένα προσωπικό το οποίο να είναι απόλυτα δεσμευμένο, το οποίο το έχουμε, δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα όσον αφορά την διαφάνεια. Έχουμε στα πλαίσια του ECDC δικούς μας εμπειρογνώμονες, γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους, είναι πραγματικοί επαΐοντες στον τομέα τους και έχουμε δημοσιεύσει τη δική τους δήλωση συμφερόντων. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση λοιπόν συμφερόντων, όλα είναι διαφανή στην ιστοσελίδα μας. Και ορισμένοι εμπειρογνώμονες είχαν συμβουλευτικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κάποιοι εξωτερικοί δηλαδή εμπειρογνώμονες. Τα περισσότερα πράγματα όμως, περισσότερες εξολογήσεις γίνανε από δικούς μας δεν υπήρχαν κάποιες διασυνδέσεις ύποπτες με φαρμακευτικές εταιρείες. Για τους πρασίνους... Ευχαριστώ. Εκτίμησα ιδιαίτερα κυρία Τεστόρη αυτή την βούληση που, λέτε, που έχετε για να, και μιλάτε για πολιτική βούληση αλλά για να έχουμε μία αλληλέγγυα Ευρώπη αγορά, αγορά κοινή αγορά εμβολίων κτλ πρέπει να είναι αξιόπιστη η Ευρώπη άκουσα την κυρία Ντεπάζ η οποία λέει να σταματήσουμε τον πόλεμο συμφερόντων ο κύριος Σπρίγκερ λέει ότι έχει πολύ καλούς εμπειρογνώμονες ωραία και λέει ότι το ΣΕΝΤΕΣΕ χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε επίπεδο των ΜΑ είναι πολύ πιο λεπτό το θέμα γιατί χρηματοδοτούνται ε, το, το μεγαλύτερο βαθμό από τα, φαρμα, τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και έχουμε εδώ λοιπόν και διαπιστώνουμε μάλλον από τις εφημερίδες ότι μέλη του ΜΑ συμμετείχαν στην έγκριση για το ταμιφλού ενώ ταυτόχρονα εξαρτώντα σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα εργαστήρια. Λοιπόν, πρέπει να αποφύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή να μην έχουμε στο MA τους ε, όσους εργάζονται για φαρμακευτικές εταιρείε. Ευθύνες λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβετε ότι οι επιστημονικές επιτροπές είναι ανεξάρτητες και η βασική τους ευθύνη να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για να λειτουργήσει η Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη όμως είναι αυτά τα οποία διορίζουν τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή ή στις Επιτροπές, οι οποίες ε, δεν σχετίζονται με καμία χρηματοδότηση, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ουσιαστικά από τις φαρμακευτικές εταιρείες, ακόμα και να αυτές καταβάλουν 80% των κονδυλίων λειτουργίας των ε, Επιτροπών. Υπάρχει σαφής παρακολούθηση προκειμένου να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και ήδη σήμερα αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό στα πλαίσια της ε, Επιτροπής. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία επίδραση στις επιστημονικές επιτροπές από το σύστημα χρηματοδότησης. Λειτουργούν οι επιστημονικές αυτές επιτροπές ανεξάρτητα από το σύστημα χρηματοδότησης. Επίσης, όταν η Επιτροπή γνωμοδοτεί, δεν μπορεί κανένα κράτος μέλος να επηρεάσει τη γνωμοδότηση αυτή ακριβώς επειδή υπάρχει απαραίτητη εξακρίβωση, επαλήθευση της ποιότητας. Έχουμε, όπως σας είπα, ένα σύστημα αξιολόγηση ομοτήμων, υποβολής εκθέσεων από εισηγητής, από εισηγητές, επαλήθευση αφός, από συνεισηγητές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τελική γνωμοδότηση είναι απολύτω απολύτως ανεξάρτητη και κανένα κράτος μέλος δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει οποιαδήποτε απόφαση. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσω. Donc, je Λοιπόν, σας παίρνω τις μετρητές αυτά τα οποία λέτε. Θα έχουμε λοιπόν τότε δηλώσεις ε, συμφερόντων. Πρέπει λοιπόν όσοι αναλαμβάνουν ευθύνες να είναι εντελώς έξω από τα φαρμακευ... τις φαρμακευτικές εταιρείες. και μπορείτε να παρέχετε και τις ε, κλινικές ε, μελέτες για τη χορήγηση αδειών ε, κυκλοφορίας των φαρμάκων όταν εσείς δεν βγάζετε αυτά τα φάρμακα στην αγορά. Όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τα στοιχεία αυτά διατίθενται στο διαδίκτυο. Μπορώ να σας δείξω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και η δεύτερη ερώτηση. η πρόσβαση στα έγγραφα. Δημοσιεύουμε στην αξιολόγηση τα στοιχεία αυτά τα οποία διατίθενται μετά την αδειοδότηση και κατόπιν αιτήματος εταιριών ή και ιδιωτών θα μπορέσουμε να αντιθέσουμε τέτοια στοιχεία, άρα να καταλάβετε ότι ο όγκος πληροφοριών που έχουμε είναι τεράστιος. Μιλάμε για εκατομμύρια έγγραφα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άμεση πρόσβαση. Είναι τεχνικής φύσης το πρόβλημα. Και θα προτείνουμε την Πέμπτη στο Διοικητικό Συμβούλιο μια νέα πολιτική για την πρόσβαση στα έγγραφα και θα προτείνουμε τη δημοσίευση όλων των κλινικών ε, στοιχείων από τις ε, κλινικές έρευνες. Ευχαριστώ κύριε Ντελής. Θα ήθελα να πω το εξής. Η δημόσια πρόσβαση ρυθμίζεται από την νομοθεσία για την έγκριση για την αγορά και μόνο οι παιδιατρικές εγκύκλοι κατόπιν αιτήματος ε, του Κοινοβουλίου διατήθηκαν, ετέθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εάν εξετάζει τις σχετικές οδηγίες. Άρα θα, κληθεί, θα κληθείτε κι εσείς να αποφασίσετε και να καθορίσετε ποια είναι το ποιο επίπεδο ε, πρόσβασης του κοινού στα κλινικά στοιχεία. Αυτό όμως ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Δεν εξαρτάται από κάθε μεμονωμένη υπηρεσία. Η κυρία Ματία, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Eh, ναι, Πρόεδρε. Ήθελα να επιμείνω και να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο για να, για να διδαχτούμε από την κατάσταση που βιώσαμε στο παρελθόν και χαίρομαι επίσης που γίνεται μία απόπειρα να δημιουργηθεί ένα νέο πρωτόκολλο για τα κλινικά τεστ, όπως επίσης και για το θέμα των κοινοτικών αποθεμάτων. Πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτά τα αποθέματα. Αλλά όμως ε, υπάρχει ένα πρόβλημα για τη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε ακόμα. Ρωτώ, Πώς σκοπεύετε εσείς να ανακτήσετε την αξιοπιστία σας άμα συμβεί πάλι κάτι αντίστοιχο στο μέλλον και μετά από όλα όσα συνέβη κατά τεράστια λάθη και η έλλειψη επικοινωνίας δεν, έχει να, δεν έχουν να κάνουν με τα διάφορα ονόματα τα οποία δόθηκαν στην πανδημία. Άμα έχουμε εμείς σε μία νέα αντίστοιχη κατάσταση, έχουμε διαπιστώσει ποια είναι, ποιες είναι οι διάφορες ομάδες, αν αρνηθούν ας πούμε οι ομάδες κινδύνου να, να, να, να, εμβολιαστούν, τι κάνουμε. Η διαφάνεια και πώς θα την ε, εξασφαλίσουμε για το μέλλον. Ο κύριος Πρέγγερ, θα ήθελα να σχολιάσω. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα της ε, εμπιστοσύνης του κοινού. Αυτό δεν άπτεται μόνο ε, της γρήπης αλλά και του ιού του παπιλώμα αφορά όλα τα συστήματα και τα σχέδια εμβολιασμού και των παιδικών ασθενειών. Μου ζητήθηκε από την Επιτροπή Αναθεώρησης της Γενέβη και είμαι πεπισμένος ότι και η ΠΟΗ κατανοεί ότι αν ε, ανακηρύξουμε την φάση 6 της πανδημίας, τότε οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν να μιλάνε για την ισπανική γρήπη κτλ. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η λέξη πανδημία, γιατί έχει λάθος, δεν είναι λάθος εντυπώσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί αν υπάρξει ένας νέος ιός και γι' αυτό λοιπόν ζητώ πιο πολύ έρευνα για να είναι καλύτερη η αξιολόγηση, η πρόβλεψη του μέλλοντος. Και εδώ το ECDC θέλει να δραματίσει το ρόλο του και να λάβει τις ευθύνε του. Γιατί εμένα με ανησυχούν. Με ανησυχεί το θέμα της εμπιστοσύνης του κοινού. Ευχαριστώ, Ζιλ Πανιό. Δύο λόγια. Για να σας πω πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα θέματα για την καθημερινή μας ζωή. Χαίρομαι ιδιαίτερα να όταν διαπιστώνω ότι υπάρχει πολιτική βούληση ε, και νομική βάση. Συμφωνώ βέβαια με την Τάγμαρ ότι η νομική βάση δεν φτάνει μου από μονάχη της. Θα πρέπει μετά το Συμβούλιο να εφαρμόσει μία ευρωπαϊκή πολιτική. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια κοινοτική πολιτική για ένα θέμα σαν και αυτό. Εσείς λοιπόν πέρα από τις ε, καλές ε, προθέσεις ε, του κυρίου Ράιντερς ή της Σουηδικής Προεδρίας θα πρέπει να αναλάβετε ένα ρόλο πρωτοπορίας. Και αυτό και λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή και όλο αυτό το φιάσκο, την καχυποψία, την αναξιοπιστία που είναι πολλά πράγματα που συσσωρεύονται ως αισθήματα του κοινού απέναντι στα ευρωπαϊκά όργανα. Τι θα, γι, τι, θα γίνει τώρα στις 5-6 Οκτωβρίου. Καταφθάνει η γρήπη λόγω του χειμώνα που καταφθάνει επίσης και μου είπαν ότι υπάρχει ένα εμβόλιο που θα μας επιτρέψει να, να ε, είμαστε καλυμμένοι όχι μόνο για την κανονική γρήπη του χειμώνα, αλλά και για την γρήπη H1. Η κυρία Τεστόρη, για τα ζώα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τον εμβολιασμό που αγοράζει τα εμβόλια που ορίζει ποια τμήμα της Ευρώπης θα πρέπει να εμβολιαστούν και πόσα ζώα θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αυτό λοιπόν δεν είναι αμφιλεγόμενο. Τα κρατημέλη επακούν γιατί υπάρχει νομική βάση επί σειρά ετών. Θεωρώ λοιπόν ότι στον τομέα της δημόσιας υγείας βρισκόμαστε στις απαρχές. Κάποια στιγμή θα καταλήξουμε και εμείς εκεί. Και για τα εμβόλια θα δώσω το λόγο στον Τόμας. Α, όχι. Δεν ξέρει δεν ξέρω κατά πόσο ποια είναι το πεδίο εφαρμογή του νέου εμβολίου για τη νέα γρήπη και για τα νέα φάρμακα. Το νέο εμβόλιο έχει συσταθεί από την ΠΟΗ και έχει ξεκινήσει να χορηγείται Και θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουμε τα στελέχη και για την εποχιακή γρήπη. Θα δούμε κατά πόσο θα είναι τετραδύναμο ή τριδύναμο το εμβόλιο. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία που ακολουθείται κάθε έτος. Η κυρία Παράνοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι επειδή όλα αυτά συμβαίνουν για δεύτερη φορά, γιατί πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια έχουν εξοδευτεί και αυτά τα χρήματα δεν χρησιμεύσαν ιδιαίτερα. Έχω λοιπόν μία πρόταση και επειδή εδώ όλοι οι φορείς αναφέρουν ότι τα πήγαν καλά, εγώ πρέπει να πω ότι δεν με ικανοποίησαν οι απαντήσεις τους θεωρώ ότι καλά τα πήγαν τα ανέφεραν τι θα κάνουν στο μέλλον. Θα προτείνω να ζητήσουμε από τη Γενική Διεύθυνση να υποβάλει σχέδια ελέγχου για την ΕΜΕΑ και το ECDC και να ζητήσει από το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει εκθέσεις για την απόδοσή τους μεταξύ 2007 και 2010 και αυτά να γίνουν στο μέλλον συγγνώμη, προκειμένου να μην έχουμε στο μέλλον μία γρήπη των ψαριών. Δεν ξέρω κι εγώ πώς θα αποκαλείται αυτό και ζητώ και συνεργασία με την Επιτροπή μας. Mr. Lundgren. I could ensure you that we are... Μα σας διαβεβαιώ ότι όντως υπάρχει μια εσωτερική υπηρεσία ελέγχου Έχουμε επίση και τι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και το λεκτικό συνέδριο που κάνουν συστηματικού ελέγχου σε όλε τι διαδικασίε μα, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε την πανδημία. Επομένω, ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη πάρα πολλοί έλεγχοι όσον αφορά την απόδοση τη δική μου υπηρεσία. Το δέχομαι αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε να γίνει κάποιο ειδικό ξεχωριστό τώρα έλεγχο για την πανδημία τη γρήπη, τότε α γίνει. ο κύριος Σπρέγγερ, ούτε κι εγώ έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα έρχεται το λεκτικό συνέδριο να μας επισκεφθεί στο ECDC, επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κυρία Ρομπέρ και η κυρία Τεστόρη ουσιαστικά έχουν ε, τονίσει τον πυρήνα το του προβλήματος δεν ε, μιλάμε στον αέρα. Και εδώ στο Κοινοβούλιο το 2006 εγκρίναμε μία ε, έκθεση του, Αδάμου, του κ. Αδάμου, μία έκθεση πρωτοβουλίας με ένα ολόκληρο σενάριο σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Κοίταξα το ψήφισμα. Ήταν ένα ψήφισμα 47 παραγράφων. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό το έργο. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό το έργο του κυρίου Αδάμου. Αλλά να ρωτήσω την κυρία Τεστόρη. Το γνωρίζετε το έγγραφο αυτό. Και όλες τις συστάσεις που έκανε τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι εξακολουθούν να είναι πολύ επίκαιρες και θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν ιδιαίτερα. Τα κοιτάξατε αυτά. Κοιτάξατε, ελέγξατε κατά πόσον έχει εφαρμοστεί κάτι από όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά τεράστιο το καθήκον αυτό που ε, απευθύνεται και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 48 συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα εξέτασε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι έκανε με τις συστάσεις αυτές. Sure, you know, Εννοείται, ασφαλώς. Θα πρέπει να σε ομολογήσω ότι εγώ προσωπικά δεν τα έχω μελετήσει, αλλά σίγουρα τα έχουν μελετήσει οι υπάλληλοι μας. Έχουμε και εμείς ε, δημοσιεύσει τέτοιες αναθεωρήσεις. Εννοείται λοιπόν ότι έχουμε κοιτάξει τις συστάσεις αυτές. Από αυτά προκύπτει η πολιτική μας άλλωστε. Ο κύριος Βελμούτ ο Η κυρία Βελμούτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που υπόθηκαν και έχουν εν μέρει απαντηθεί τα ερωτήματά μου γιατί άπτονται της διαφάνειας και τις σχέσεις που υπάρχει με τις φαρμακευτικές εταιρείες για την μελέτη. Άκουσα όσα μας είπαν από την ΕΜΑ και από το ECDC. Επειδή είναι εδώ η κυρία Γιάκα, να ρωτήσω γιατί δεν μπορούν να γίνουν αυτά και για την ΠΟΗ, γιατί αν καταλαβαίνω σωστά, μάλλον καταλαβαίνω ποια είναι η σχέση μας με την ΠΟΗ, αλλά ακολουθήσαμε τη σύσταση να περάσουμε στο επίπεδο συναγερμού 6. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν αυτές οι πληροφορίες και νομίζω ότι είναι πραγματικά μεγάλη ντροπή που δεν υπάρχει διαφάνεια στον τομέα αυτό. Η ε, κυρία Γιάκοπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω παρά το γεγονός ότι δεν είμαι μέλος του πάνελ αυτού. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η Επιτροπή Κατεπηγόντων είναι αυτή που συστήνει το γενικό, στον Διευθυντή σχετικά με το επίπεδο της ε, ετοιμότητας της και ακολουθήσαμε τις συστάσεις λοιπόν αυτής της Επιτροπής. Ο λόγος ήταν να αποφευθούν οι πολιτικές εντάσεις και η άσκηση πολιτικής πίεσης και πίεσης από τις φαρμακευτικές ε, εταιρείες. Γι' αυτό λοιπόν εσωτερικά αποφασίστηκε να μην δημοσιεύτουν τα στοιχεία αυτά παρά μόνο στο τέλος. Ο τώρα που ανακηρύχθηκε η λήξη της πανδημίας, τίθεται το θέμα της σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Ωστόσο, σημειώνουμε το μήνυμά σας και ως μήμα της ε, διαδικασίας αναθεώρησης θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο είναι πρόκειται η σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα διαφανείς και αυτό το μετέφερα και στην ΠΟΗ, γιατί πρόκειται για μία από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι χρειαζόμαστε πάντα διαφάνεια σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Και η σύστασή μου είναι να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στην προκειμένη περίπτωση. Και είμαι βέβαιη ότι θα το αναθεωρήσουμε αυτό και στη σχετική επιστροπή του ΣΠΟΗ. intervenir tout à l'heure euh, certains de nos collègues όταν ορισμένοι συνάδελφοι εξέφραζαν καχυποψία για το τι ε, συνέβαινε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ήθελα να πάρω το λόγο για να πω απλώς το εξής, ότι εμείς είμαστε αυτοί που ελέγχουμε ετησίως αυτούς τους οργανισμούς. Έχουμε, ελέγχουμε μόνιμα ε, τους ε, οργανισμούς μας και ΜΕΑ είναι ε, μία από τις καλύτερες, ένας από τους καλύτερους οργανισμούς. Σταματήστε λοιπόν όλες αυτές τις τύρες ε, παρατηρήσεις γιατί όλα είναι ελέγξιμα. Πρόκειται για ένα συμπλήρωμα πληροφόρησης διότι σοκάρομαι πολλές φορές ακούγοντας μερικά πράγματα. Μάλιστα, Ελίντα Μακέβεν. Σας ευχαριστώ. Το ζήτημα αυτό της προμήθειας και των συμβάσεων προμήθειας των εμβολίων. Θα ήθελα να το δούμε λίγο περισσότερο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με νέο κοινό τρόπο. Επίσης, ε, ποια είναι η τιμή που κατέβαλαν τα κράτη-μέλη για τα εμβόλια. Ορισμένα κράτη-μέλη πλήρωσαν περισσότερα από κάποια άλλα και δεν κατάφεραν να πάρουν τα εμβόλια τα οποία απαιτούσαν. Ποιος έλαβε λοιπόν τα εμβόλια στην κάθε χώρα πώς έγινε η κατανομή, θα έπρεπε ουσιαστικά το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί στη νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι αν είχαμε καταφέρει να εξοικονομήσουμε χρήματα, θα είχαμε και μια καλύτερη πολιτική συμβάσεων όσον αφορά την προμήθεια των εμβολίων. Ο κύριος Ράιν, να θέσω και εγώ ένα ερώτημα. Υπάρχουν σχέδια για την υποστήριξη χωρών που δεν κατάφεραν να βρουν εμβόλια. Υπάρχει δηλαδή κάποιο σημείο αλληλεγγύης. Στι 13 ε, Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση όσον αφορά το ζήτημα αυτό των συμβάσεων. Σε συμπεράσμα του Συμβουλίου μα ζητήθηκε να εξετάσουμε διαφορετικέ συναλλακτικέ. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προετοιμάσει ήδη ένα έγγραφο το οποίο αναλύει τι διαφορετικέ ε, επιλογέ δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το ε, αρμόδιο δίκαιο των συμβάσεων και έγινε και μία συνάντηση την προηγούμενη Παρασκευή όπου συζητήθηκε το έγγραφο αυτό προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να δουν τα θετικά και τα αρνητικά κάθε εναλλακτική λύση. Προβλέπεται τώρα μία νέα συνάντηση στα τέλη Οκτωβρίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί το έγγραφο και προκειμένου να υποβληθεί στην Επιτροπή Υγείας στις αρχές σε Δεκεμβρίου, σε 7 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα. Ουσιαστικά τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν το έγγραφο αυτό, να κάνουν μια πολύ καλή ανάλυση των νομικών επιλογών που υπάρχουν όσον αφορά αυτόν τον προτινόμενο συνδυασμό κοινών δημοσίων συμβάσεων και να ληφθεί κατά αυτόν τον τρόπο μια απόφαση το Δεκέμβριο όσον αφορά τις διαφορετικές τιμές. Σαφώς υπήρχαν διαφορετικές τιμές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, αλλά αυτό εξαρτάται από το αν είχαν πρώτερες συμφωνίες αγοράς για κάποια εμβόλια, αν είχαν συνάψει τα ίδια συμβολίες του 2008-2009. Αυτό όμως είχε να κάνει και με τον αριθμό των πολιτών που προτίθονταν να εμβολιάσουν. Ποιες ήταν οι συνθήκες μεταφοράς και παράδοσης. Ποιες ήταν οι συνθήκες ε, ανάληψης ευθύνης. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί παράγοντε επηρέαζαν τη διαμόρφωση των τιμών και γι' αυτό το λόγο οι τιμέ ήταν διαφορετικέ από τη μία χώρα στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μία πρόταση προκειμένου να υπάρχει μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση των τιμών, των όρων, των συνθήκων καθώ επίση και των άλλων συνθήκων των συμβατικών για την παράδοση των εμβολίων. Καρίν Κάμπερ. Η Λίντα υπήρξε έλλειψη ε, εμβολίων τότε, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να αγοράσουν εμβόλια και δεν μπορούσαν. Ναι, αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν νωρίτερα, ότι κάποια κράτη-μέλη ε, δεν είχαν ε, συμφωνίες αγορών αγοράς για εμβόλια. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς προσπάθησε να οργανώσει μια ένα κοινό διαγωνισμό για τέτοιες συμβάσεις βάσει των εμπειριών που είχαμε αποκτήσει και από άλλες χώρες και κατά δεύτερον διοργανώσαμε ένα σύστημα μεταφορών με μεταξύ χωρών που είχαν υπερβολικό αριθμό εμβολίων και των χωρών που είχαν έλλειψη. Αυτές ήταν οι πρωτοβουλίες που είχαμε λάβει το φθινόπωρο του 2009. Ελπίζουμε να διδαχτούμε από τις εμπειρίες αυτές και να ξεκινήσουμε καινούργιες πρωτοβουλίε πλέον. Ε, I'm sorry, I'm taking the, ναι, συγγνώμη που παίρνω το λόγο τώρα. Δεν είμαι στο σωστό πανέλ, αλλά θα ήθελα να μιλήσω για την πολιτική δέσμευση των Υπουργών. Να σας υπενθυμίσω ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2009 οι Υπουργοί ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουν τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Ζήτησαν από την Επιτροπή το 2009 ήδη να κάνουν μια ει ανάλυση. Όλοι οι Υπουργοί το ζήτησαν αυτά τον Οκτώβριο του 2009. Next speaker is Karin Kallenbach. Η επόμενη ομιλητρία. Μία ερώτηση προς τον ε, διευθυντή Σπρέγγερ, ο οποίος, ήταν άμεσος, ο οποίος δεν ήταν άμεσα ε, ενδιαφερόμενος, αλλά το έθιξε το θέμα αυτό στις εισηγήσεις του. Θεωρώ ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας οδήγησαν στην μείωση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά κράτη-μέλη διαπιστώσαμε ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις παιδικές ασθένειες περιορίζονται οι εμβολιασμοί. Αναμένεται λοιπόν πραγματικά ε, πανδημίες, υπάρχουν προφυλάξεις στα κράτη-μέλη προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τέτοια ζητήματα. Thank uh, uh, Σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένα λόμπι κατά των εμβολιασμών και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Γιατί τρομάζουν τον κόσμο χωρίς στοιχεία. Επίσης, να τονίσω το εξής. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια νομική πτυχή, αλλά τελικά εξαρτάται και από τον πολίτη που πάει στο γιατρό. Αν ο γιατρό δεν είναι πεπισμένο ότι χρειάζεται ο εμβολιασμό, αν ο γιατρό δεν κατανοεί την ανάγκη αυτή, υπάρχει πρόβλημα και χαίρομαι που στις 16 Νοεμβρίου έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα αντιβιωτικά. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια λυσίδα επικοινωνίας μέσω των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Προσπαθούμε να πείσουμε του γιατρούς ότι είναι σημαντικό να μειωθεί να μειωθεί η χρήση των ε, αντιβιωτικών. Ελπίζω του χρόνου να υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά της γρήπης. Και να δώσουμε επίκεντρο να υπογραμμίσουμε και τη σημασία των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Euh, euh, ήθελα, θα ήθελα να να συνεχίσουμε όλη αυτή τη συζήτηση μεταξύ κρατών μελών και κομισιών για όλη αυτή την ιστορία των εργαστηρίων που για τους ε, που για τις αντεδείξεις των ε, φαρμάκων τις ευθύνες τις φέρουν τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας? Ότι ότι όλες τις παρενέργειες τις δείχνουν στην πλάτη των κρατών μελών. Ας πούμε η ναρκοληψία πώς βγήκε στη φόρα από τις εθνικές αρχές της Σουηδίας, μετά από τη Φιλανδία και μετά από το ΕΜΑ. Αν είναι υπεύθυνο το ΕΜΑ για το θέμα των παρενεργειών, τι κάνετε και πώς το ΣΕΝΤΕΣΕ προχωρά στη σύνταξη μελετών για να διαπιστώσει τόση ότι πρόκειται για παρενέργειες που οφείλονται στον εμβολιασμό και όπου πλήττονται κυρίως τα παιδιά. Ποιος θα απαντήσει, ο κύριος Σπρέγκερ και η κυρία Τεστόρη. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων βρίσκεται σε ηγετική θέση όσον αφορά την ανάλυση των παρενεργειών, αλλά και το ECDC ασχολείται πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό, γιατί δεν είμαστε απεπισμένοι ότι πρόκειται πράγματι για παρενέργειες του εμβολίου. Στεργαζόμαστε πάντως με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και κάνουμε συγκεκριμένες μελέτες. Εξετάζουμε κάποιες πραγματικές περιπτώσεις παρενεργειών και τις συγκρίνουμε με διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν έχουν εντοπιστεί παρενέργειες αυτές. Θα θέλαμε πραγματικά να εντοπίσουμε τους λόγους των φαινομένων αυτών. Πρόκειται για πραγματικό φαινόμενο και πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στους πολίτες. Αν τελικά οι παρενέργειες αυτές δεν συνδυάζονται με το εμβόλιο, γιατί και αυτή η πιθανότητα υπάρχει. Να επιβεβαιώσω κι εγώ ότι ασχολούμαστε με το ζήτημα αυτό, ότι έχουμε συλλέξει τις περιπτώσεις αυτές στη βάση δεδομένων μας και ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση αυτή τη στιγμή ότι αυτές οι παρενέργειες συνδέονται με το εμβόλιο. Ξεκινήσαμε πάντως μια διαδικασία εξέταση του φαινομένου σε συνεργασία με το ECDC και με άλλες υπηρεσίες. Ξεκινήσαμε συγκεκριμένα μελέτες που θα μας επιτρέψουν να εξακριβώσουμε αν όντως υπάρχει συσχέτιση με το εμβόλιο ή αν υπάρχει κάποια άλλη συσχέτιση δηλαδή με την ίδια τη γρήπη, με τον ίδιο τον ιό, με την ίδια τη μόλυνση. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιος ε, συσχετισμός με την συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας. Ελπίζουμε ότι στις αρχές του 2011 θα έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα από τις μελέτες μας αυτές. Το θέμα της ευθύνης για τις παρενέργειες στο ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι και λέει ότι είναι υπεύθυνη η βιομηχανία. Στο πλαίσιο λοιπόν της χορήγησης άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου και στα πλαίσια των πληροφοριών που δίνονται για τις παρενέργειες και που επικυρώνονται κατά τη χορήγηση της άδειας. Αν ξεπερνάνε λοιπόν αυτές οι παρενέργειες το επιτρεπόμενο όριο, στη βάση της χορήγησης της άδεια, τότε η βιομηχανία είναι υπεύθυνη. Ευτυχώς ε, δεν είχαμε... Ε, δεν μας δόθηκε ευτυχώς η ευκαιρία να αναρωτηθούμε και να προβληματιστούμε για το πρόβλημα. Τι θα συνέβαινε δηλαδή αν το κράτος μέλος με τη φαρμακευτική εταιρεία είχε ένα δικό του, ε, ένα δικό του συμβόλαιο με τη φαρμακευτική εταιρεία, τι θα γινόταν με την ευθύνη, θα ίσχυε, ε, θα ίσχυε η η διάταξη του κανονισμού και κυρία Λεπάζ σε εσάς ρωτάω που είστε διάσημοι νομικός πρώτη φορά μας έτυχε τέτοιου είδους ε, επεισόδιο. <coughs> Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν είναι υπεύθυνη η φαρμακευτική εταιρεία για οποιαδήποτε παρενέργεια η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Με αυτήν η γνώμη μου άλλοι μπορεί να, ως νομικός, άλλοι μπορεί να έχουν άλλες γνώμες. Πάολα στο μελλοντικό κανονισμό πρέπει να ληφθεί υπόψη το θέμα της ευθύνης. Μάλιστα κύριε Τεστόρη, είναι σαφές ότι το ερώτημα αυτό, το ζήτημα αυτό της, ε, των πανεργειών συμπεριλαμβάνεται στις συζητήσεις μας, τις τρέχουσες. Και θα πρέπει να πω σε ό,τι το παρελθόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, πρόσβαση σε όλες τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των κρατών μελών και από τα κρατημέλη γιατί πολλά κρατημέλη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Αλλά είναι σαφές ότι βάσει των πέντε που έχουμε στη διάθεσή μας θα συμπεριλάβουμε τα στοιχεία αυτά στο μέλλον. Νομίζω ότι ήταν ο δεύτερος γύρος των ερωτών απαντήσαν αυτός. Πολλά ενδιαφέροντα ακούσαμε και τώρα έχουμε δύο συνεισηγητές, τον κύριο Πέτρελε και τον, την κυρία Βέλμοντ, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο προτού η Μισελ κάνει τα τελευταία σχόλια, τα τελικά σχόλια. Λοιπόν, στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν συνάδελφοι που δεν είναι απαραίτητα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, διότι εμείς θέλουμε να εμπλέξουμε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται και που μπορεί να είναι χρήσιμοι στην Επιτροπή μας. Οι κριτικές ε, και τα ερωτήματα ε, για την πανδημία ε, προέκυψαν πρώτα από τους ίδιους τους εμπειρογνώμονες και μετά πέρασε στην κοινή γνώμη. Και εμείς, περάσαμε, πε, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ακούμε τους πολίτες και οι πολίτες είχαν πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με το πώς λειτουργήσε ο εμβολιασμός. Για παράδειγμα ορισμένοι αναρωτήθηκαν πώς ε, πώ ε, λειτουργήσε ο εμβολιασμό. Ορισμένοι γιατροί, οι γιατροί εμβόλιασαν τον κοσμάκι, αλλά ορισμένοι γιατροί δεν θέλησαν να εμβολιάσουν του εαυτού του. Και μερικοί αναρωτήθηκαν τι, τι δημιουργήθηκε πρώτα, η γρήπη ή το εμβόλιο. Μας λείπουν πολλές φορές τα χρήματα, όχι μόνο για την πρόληψη αλλά και για τη θεραπεία. Και η κατάσταση συνεχώς υποβαθμίζεται και σίγουρα θα μπορούσαμε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε άλλες πανδημίες. Πρέπει λοιπόν εμείς να θεσπίσουμε έναν κανόνα, να μην τρέχουμε, να μην ξοδεύουμε πολύ, να μην σπαταλάμε χρόνο. Πρέπει όμως να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε, μία, σε έναν ορισμό και καταπολέμηση των πανδημιών με επιστημονικά κριτήρια. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Υπήρξαν αμφιβολίες που εκφράστηκαν Ορισμένοι έχουν, τις έχουν ακόμα. Ακούσαμε τι είπε η ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμείς ως κράτη-μέλη θα πρέπει να προσέξουμε και τις προηγούμενες φάσεις της πανδημίας. Η Κομισιόν μας είπε ότι εργάζεται για μία νέα νομική βάση. Σίγουρα χρειάζεται πολιτική βούληση να παράβα το τέτοιο. Εμείς οι βουλευτές ενδιαφερόμαστε Εμείς λοιπόν πρέπει να ενημερωνόμαστε. Πολλοί οργανισμοί από μόνοι τους αποφάσισαν να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θέλουμε να υπάρχει συμφερόντων, δεν θέλουμε να υπάρχει συμβατότητα, δεν θέλουμε να υπάρχει προσβολή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Να δούμε λοιπόν στο μέλλον πώς θα εμβαθύνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πέτρελα. Η κυρία Βελμότα, ευχαριστούμε πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το εργαστήριο του σημερινό και θα ήθελα να πω ότι προφανώς ε, αμφισβητούμε τον μεγάλο αριθμό εμβολίων που αγοράστηκαν. Το θέμα όμως είναι ότι και τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε αγοράσει τα εμβόλια αυτά ως ε, πολίτες. Αναμένουμε και θέλουμε οι δημόσιες αρχές να είναι προετοιμασμένες για περίπτωση κρίσης και θα είναι μεγάλη κριτική που θα δεχόμασταν αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια. Ωστόσο, Υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν σήμερα σε ό,τι αφορά την ε, διαφάνεια, σε ό,τι αφορά τους εμπειρογνώμονες, τα ειδικά συμφέροντα και νομίζω ότι πολλές ε, ιδέες ακούσαμε και πολλά στοιχεία λάβαμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας εδώ στην Επιτροπή μας. Λογικό μου φαίνεται σε μελλοντικές πανδημίες να υπάρχει μια κοινή διαδικασία δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα μας ενίσχυε και θα βελτίωνε τις ε, όρους για τα κράτη-μέλη, το οποίο είναι ενδιαφέρον και για τα μικρά τα κράτη-μέλη ιδιαιτέρως. Θα δούμε ποιες προτάσεις θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μάθαμε από τα διδάγματα του παρελθόντος, προκειμένου στο μέλλον να είναι πιο διαφανή και πιο αποτελεσματική η διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και ε, είμαι αισιόδοξη ότι αυτό θα συμβεί. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ριβαζή θα πρέπει να τα α, συνενώσει όλα αυτά σε μία έκθεση, να της δώσω το λόγο για να ολοκληρώσει. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σήμερα. Μεγάλο ευχαριστώ, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Είχαμε μία ερευνητική επιτροπή στη Γαλλία 90 εκατομμύρια δόσεις ε, παρασκευάσαμε στην ε, Γαλλία για τη διαχείριση της ε, γρήπης. Ξοδέψαμε τα περισσότερα λεφτά. Είχαμε στη Γερουσία λοιπόν μια ερευνητική επιτροπή και μετά είχαμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Να σας διαβάσω κάτι που λέει η έκθεση. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκε, έγινε η διαχείριση της γρήπης όχι μόνο από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο είναι ανησυχητικό. Διότι ορισμένες συμβουλές οι οποίες δόθηκαν και αποφάσεις που δόθηκαν ε, ε, οδήγησαν σε μία στρέβλωση των στόχων των υπηρεσιών δημόσιας υγείας ανά την Ευρώπη από προσανατόλισαν την Ευρώπη από τους στόχους δημοσίας υγείας και τους πολίτες. Αυτή ήταν η διαπίστωση και όπως έλεγε και ο συνάδελφος τελικά ο κόσμος δεν έχει πια εμπιστοσύνη. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας θα πρέπει να βοηθήσει ούτω ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίος πολίτης. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αν θέλετε να προχωρήσουμε πρέπει να αναλύσουμε το παρελθόν για να μπορέσουμε να δούμε πού δυσλειτουργήσαμε. Αλλά όλα αυτά επικοδομητικά. Δεν το βλέπουμε καταστροφικά το θέμα. Δεν θέλουμε απλώς να είμαστε έρμεα κριτικής και δεν θέλουμε ο κόσμος να λέει ορίστε η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη η οποία οικοδομείται, η οποία είναι αλληλέγγυα, η οποία ψάχνεται και η οποία έχει εμπειρογνώμονες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα προχώρημα των διεθνών, διεθνών οργανώσεων. Δεν, δεν αποτελούν τους ουραγούς. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και τι πρέπει να ξαναδούμε τι εστί πανδημία. Δεν μπορείτε να αφήνετε την πανδημία μόνη της να λέει ότι η πανδημία είναι θέμα γεωγραφικής ε, επέκτασης. Ε, όχι. Εμείς πρέπει να πούμε ότι διαφωνούμε. Και είτε εσείς θα το παλέψετε το θέμα στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας διότι συμμετέχει εκεί η Κομισιόν ή αλλιώς θα πρέπει εμείς ευρωπαϊκό επίπεδο να ορίσουμε περί τίνος πρόκειται. Επίσης άκουσα να μιλάμε για ευελιξία και ανεξαρτησία. Ωραία. Καλύτερη αξιολόγηση των ρίσκων. Μα αυτό είναι απαραίτητο διότι αλλιώς ε, θα, θα, θα ξαναπέσουμε αύριο μεθαύριο σε μια άλλη πανδημία. Αν δεν αρχίσουμε να θα λίγο, τελικά ο κόσμος δεν θα πάει να εμβολιαστεί. Δεν είναι θέμα ποιος είναι υπέρ ή κατά του εμβολιασμού. Αλλά θα λέει ο κόσμος ότι σε τι χρειάζεται. Διότι είπαμε για τη γρήπη να εμβολιαστούν, αλλά δεν πήγανε και σχετικά με την ε, μαζική κοεμβολιασμό κατά της γρήπης, όταν υπάρχει ιός, δεν υπάρχει ιός, υπάρχει κάλυψη, 100% κάλυψη. Το δεύτερο πάνελ ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ο στόχος της έκθεσης μάλλον η έκθεση θα διαμορφωθεί και από άλλες δύο ακροάσεις που θα γίνουν για την ευθύνη, τι θα κάνει το ΣΕΝΤΕΣΕ, ποια είναι τα όρια του και οι ευθύνε του, τι μπορεί να κάνει ΕΜΑ σε επίπεδο Συμβουλίου και Κομισιόν. Να δούμε δηλαδή πού βρίσκεται η ευθύνη του, το όριο της ευθύνης του καθένα. Και η δεύτερη ακρόαση θα είναι συνεργασία με τα κράτη-μέλη, μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σήμερα το πρωί εγώ άκουσα να μιλάμε για συνεργασία. Συναντώντας τα κράτη-μέλη και τα διάφορα θεσμικά όργανα πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα. Υπ' αυτή την προπτική λοιπόν θεωρώ ότι η έκθεση πρωτοβουλίας πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε την αξιοπιστία μας και άμα υπάρξει ένας τέτοιος τρομερός ιός αύριο μεθαύριο να πούμε όλοι θα πάμε να εμβολιαστούμε και όπως είπε και η κυρία Τεστόρη δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ιστορίες όπου τα κράτη επιβαρύνονται για θέματα των εμβολιασμών. Σας ευχαριστούμε για τα συμπεράσματα αυτά. Οι τελευταίες δύο ώρες ήταν πολύ σημαντικές για τις εργασίες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Οι εκλογείς μας, οι πολίτες το κοινό περιμένει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει την κατάσταση. Και όσα συνέβησαν πέρσι, μάθαμε ωστόσο αρκετά από το εργαστήριο αυτό. Δεν είναι τίποτα θέμα. Υπήρχαν ελλείψεις, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε αυτό και θα ήταν λάθος να το κρύψουμε και θα πρέπει στο μέλλον να βελτιαστούμε, να βελτιωθούμε. Χαίρομαι που η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μας δίνει μεταξύ άλλων και μία νέα βάση. Μπορούμε πλέον να ασκούμε καλύτερο συντονισμό και μία πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα όσα ακούσαμε εδώ σήμερα. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να είναι σαφής, να είναι εμφανής ε, σε τέτοιες ε, περιπτώσεις, να μην είναι δημιουργούνται δηλαδή παρετά έξοδα, να είμαστε αναποτελεσματικοί. Πολλά ουσιαστικά ακούσαμε σήμερα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες, όλους τους προσκεκλημένους μας. Σας ευχαριστώ για την δουλειά σας, να ευχαριστήσω και την γραμματεία για την ε, διοργάνωση που δεν είναι καθόλου εύκολη της ε, σημερινής ε, συζήτησης, να ζητήσω και συγγνώμη από τους ε, πρώτους ομιλητές που ήμουν αυστηρός. Νομίζω όμως ότι ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμα τα πορίσματα του εργαστηρίου αυτού. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις μελλοντικές εργασίες και κλείνω την συνεδρίαση. On a eu des réponses. Oui. Mais la première